good morning everybody. Let's uh, start. Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση μας. Ξεκινάμε με μια ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αφρικανική Ένωση, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που τίθενται. Προγραμματίσαμε αυτήν την ακρόαση για να συνδυαστεί με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Αντίσα Μπέμπα, στην Αφρικανική Ένωση. Πρέπει να το, χρειάζεται να το αλλάξουμε όμως και θα πάμε στην Αφρικανική Ένωση. Okay. I have to speak, otherwise you don't hear. <laughs> okay. So we uh, are planning to... Λοιπόν, έλεγα ότι προγραμματίζουμε να πάμε τέλη Ιουλίου, την τελευταία εβδομάδα Τυρκουάζ πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και προετοιμάζουμε λοιπόν την επίσκεψή μας ε, για να συζητήσουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική και για να δούμε πώς έχει προχωρήσει η Αφρικανική Ένωση στην ανάπτυξη των δομών σε διάφορες χώρες. Χθες, η πρόεδρος, ε, ε, ε, Δόκτωρ Ναμίνη Τσούμα, ήταν στις Βρυξέλλες για μια μέρα μόνο Πράγμα που δείχνει ότι και εκείνοι κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν ε, καλές σχέσεις, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναντήθηκε με τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Βαν Ρόμποη. Ο πρόεδρος Σούλτς ε, ήταν ασθενής και μου ζήτησε να τη συναντήσω εγώ. Ήταν πολύ καλή αυτή η ευκαιρία γιατί έχει αναλάβει καθήκοντα από πέρυσι τον Ιούλιο και τώρα προετοιμάζει τη δουλειά τους για την 50η επέτειο της Αφρικανικής Ενώσεως φέτος και προγραμματίζουν το μέλλον για να έχουν ένα πρόγραμμα μέχρι το 2050 για τα βήματα που θα κάνει η Αφρικανική Ένωση μέχρι τότε. Συμφωνήσαμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό και για τη δουλειά που κάνει η Αφρικανική Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τη δική μας δουλειά στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να εντείνουμε τις ε, κοινέ μας συζητήσεις για να διδασκόμεθα ημένα από τους ΔΕ και να δούμε ε, τι ε, είναι αυτό που θα λειτουργήσει καλύτερα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και αυτή την οργάνωση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η ε, δόκτωρα Μίνι Τσούμα τόνισε ότι επειδή υπάρχουν πολλές βίες σειράξεις και πόλεμοι στην Αφρικανική Ένωση, καλό θα ήταν να εστιαστεί στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών σε εμπόλεμες περιοχές. Ακόμη, ε, θεωρεί χρήσιμο να οριστεί κάποιος ειδικό σύμβουλος ή συντονιστής, δεν ξέρω πώς θα ονομάσουμε αυτή τη θέση, στην Αφρικανική Ένωση, που θα ασχολείται με την σεξουαλική βία, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση λοιπόν και νομίζω ότι μπορούμε να την υποστηρίξουμε το Κοινοβούλιο δεν οφείλει να χρηματοδοτήσει τέτοιες προσπάθειες. Είναι κάτι που μπορεί να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μαζί μας έχουμε τον καθηγητή Φάλη, Και όπως βλέπετε, ε, κύριε καθηγήτα, κάνουμε ακροάσεις που δεν είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια. Είναι προσπάθειά μας ε, ε, να έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση με ακροάσεις και με συνεχή συνεργασία. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα για την ακρόασή μας και ευχαριστούμε και τις τεχνικές υπηρεσίες γι' αυτό, γιατί θα μας συνδέσουν με την δικαστή κυρία Σοφία Ακούφο από την Κάνα, πρόεδρο ε, του Αφρικανικού Δικαστηρίου για τα δικαιώματα των ανθρώπων και των λαών. Η σύνδεσή μας είναι με την Αρούσια στην Τανζανία. Σας ευχαριστούμε πολύ, ε, κυρία δικαστά Κούφο. Μας ακούτε? Σας ακούω και ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε κι εσείς. Καλή σας μέρα. Σας ακούμε και εμείς πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια ευρύτατη ημερήσια διάταξη και προσπαθούμε να δούμε πώς δουλεύουν τα θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορους περιφερειακούς θεσμούς. Θέλουμε να δούμε πώς λειτουργούν οι περιφερειακοί θεσμοί, τι έχουν επιτύχει και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν. Το κάναμε και με το ε, Αμερικανικό Δικαστήριο. Ε, χτες κάναμε μια συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους από την περιοχή ΑΣΕΑΝ και τώρα με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εσάς και περιμένουμε να μας μιλήσετε εσείς για τις εξελίξεις στο Αφρικανικό Δικαστήριο για τα δικαιώματα των ανθρώπων και των λαών. Έχετε λοιπόν το λόγο και μεταξύ αυτών που θα μας πείτε θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια και για τη δουλειά σας και αν μπορείτε να μας πείτε τι θεωρείτε ότι καλό θα ήταν να κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών καθώς και συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο λοιπόν για περίπου πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Έχω μόνο πέντε λεπτά. Έχω ήδη στείλει μια σύνοψη των όσων θα πω. Όσον αφορά το έργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Αφρικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι σωστά αυτά που έθηκα. Η, δομή των εργαλείων που έχουμε στην Αφρική τα ανθρώπινα δικαιώματα εντάσσονται στην Αφρικανική Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σύστημα προστασίας αυτών και προώθησης αυτών υφίσταται. Υπάρχει και αρμόδια επιτροπή αφρικανική. Και υπάρχουν και τα διάφορα δικαστήρια. Και το Αφρικανικό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Λαών. Το δικαστήριο επικροτεί το έργο της αρμόδιας επιτροπής Και το δικαστήριο έχει μόνο δικαιοδοσία, ε, δικαιοδοτική αρχή, εξουσία. Προσπαθεί να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά προβλέπονται στη χάρτα. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομικά. Υπάρχει σωστή ανταπόκριση. Προσφεύγουν σε εμά ε, ε, που μπορεί να είναι ή κράτος ε, ή μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Αυτοί μπορούν να προσφύγουν σε εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ποινικά θέματα. Οι εργασίες μας πλαισιώνονται από τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η δικαιοδοσία μας. Υπάρχει πρωτόκολλο αφρικανικό για τα δικαιώματα των γυναικών. Και επίση αφρικανική χάρτα για τα δικαιώματα των παιδιών. Εκεί εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο δικαιοδοσία μας.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 Uh, we Σας ακούμε, αλλά πρέπει να συγκεντρώμαστε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Από τον ήχο μέχρι τώρα σας κατάλαβα. Οι διερμηνείς όμως δεν μπορούν να καταλάβουν, σας λέει ο διερμηνέας, γιατί ο ήχος είναι πάρα πολύ κακός και δεν μπορούμε να διερμηνεύσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Can hear you. Please continue. Thank you. All right. Yes. So the the the, the so I've spoken about the challenge of this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 I think you I know that my five minutes are already up. Yes. And uh, I think maybe I will stop here. Yes. So thank you very much, uh, Justice Akufo. That was... Ευχαριστώ κυρία δικαστήνα, κυρία Ακούφο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, να βλέπουμε πόσος χρόνος χρειάστηκε για να δημιουργηθεί το δικαστήριο και τα σχέδιά σας για το μέλλον θεωρώ ότι όταν λέτε ότι υπάρχουν μόνο μερικές χώρες, έξι τον αριθμό, που έχουν αυτή τη διακήρυξη για καλύτερη, που επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση στα δικαστήρια στις ΜΚΙΟ και λέτε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός κυρώσεων του πρωτοκόλου που δημιουργεί το δικαστήριο Πρέπει να σας πω ότι εμείς όταν ασχολούμεθα με χώρες μέλη της Αφρικανικής Ενώσεως, τα ενθαρρύνουμε τα κράτη να επικυρώσουν ταχύτερα και να υποστηρίξουν με σοβαρότητα το δικαστήριο. Έχουμε τη τεχνική δυνατότητα Μπορούμε να ακούσουμε τον καθ καθηγητή Φόλα από την Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών είναι, παρακολουθεί το έργο της Αφρικανικής Ένωσης και κατά τη συζήτηση θα είχε τη δυνατότητα να παρεμβαίνετε. Καλώς. Yes. Thank you. Συμφωνεί. And, uh, I give Professor Fall... Πριν δώσω στον καθηγητή Φόλ το λόγο, καλωσορίζω και τον πρέσβη εκπρόσωπο τη Αφρικανική Ενώσεω, τον κύριο Αγιάη Καπραντέο, αν προφέρω σωστά το όνομά σα. Είστε πολύ άσχολο. Και ελπίζω να ήταν ε, αποδοτική ε, η επίσκεψη του Δ. Λαμίνη Τσούμα Ο κύριος Μαμπά Σαφόλ, ο καθηγητής Μαμπά Σαφόλ είναι εδώ. Εκπροσωπεί οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών θα παρουσιάσετε διάφορες συστάσεις. Συστάσεις Αφρικανικής Ενώσεως, Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Διαλόγου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για, το ανθρώπινο διάλο... για τα διάλογο που έγινε στην Αντίσα Μπέμπα πέρσι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, θέλετε να θέσετε διάφορα θέματα προς την Αφρικανική Ένωση. Στην Επιτροπή μας ενημερωθήκαμε και κλεισμένο των θυρών από τους ειδικού εκπροσώπους τον κύριο Λαμπρινίδη, τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα ενημέρωσε για τι συζητήσει και τα αποτελέσματα όσον αφορά τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε τα πάντα όσα γίνονται στην Αφρικανική Ένωση, να μας ενημερώσετε. Ετοιμαζόμαστε, βλέπετε, για αποστολή φέτος. Έχετε το λόγο και μετά θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις που θα υποβληθώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γέννη και την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσκληση που μου απευθύνθηκε. Απευθύνθηκε στην κοινωνία των πολιτών μέσω εμού. Ευχαριστούμε την κυρία Σοφία Κούφο, την δικαστήνα που ακούσαμε πριν για αυτά που μας είπε τη Σιχέρο που διορίστηκε επικαλή ε, του δικαστηρίου και ήταν λαμπρή παρέμβασή τη η Αφρική εδώ και περίπου 15, 18, 20 χρόνια λιγότερο από ένα τέταρτο του αιώνα η Αφρικανική Ένωση έχει θεσμικό πλωστάσιο και ε, δικαστικό δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες για αυτό το πλωστάσιο, πραγματικά πλωστάσιο ε, υπήρχαμε θεσμική αλλαγή που επιτρέπει ε, να δικάζει στην Αφρική έναν πρώην πρόεδρο της ε, Δημοκρατίας. Θα ξεκινήσει η διαδικασία στη Σενεγάλη 14 μήνες. Θα ξεκινήσει η δίκη του πρώην Προέδρου. Και αυτό χάρη σε εντολή που δόθηκε στη Σενεγάλη τον Ιούλιο του 2006 την Αφρικανική Ένωση στη Σύνοδο Κορυφής του Μπαντζούλ. Προστίθεται σε αυτό πολλά, πολλά κείμενα που θεσπίθηκαν για να σταματήσει η ατιμορρησία των σοβαρότερων εγκλημάτων στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυτή η μάχη λοιπόν, κύριοι και κυρίες βουλευτές, έχει την ύψιστη προτεραιότητα στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτά τα εγκλήματα. Άρα χρειάζεται πραγματικός πόλεμος κατά της ατιμορρησίας. όπως μου ζητήθηκε, αφού θα πάτε στην Αιθιοπία, να σας πω ότι η Αφρικανική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι λαοί πήραν μια απόφαση, ένα ψήφισμα που καταδικάζει την κυβέρνηση Αιθιοπίας. Αυτό δείχνει ότι σήμερα στην Αφρικανική Ένωση υπάρχουν φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σχετική εντολή που καταγγέλουν τέτοια πράγματα στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών. Δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα τα πράγματα όμως. Διότι η κοινωνία των πολιτών στην Αφρική δεν, αρκετά, εκπροσωπείται παρκώ στην κοινωνία των πολιτών, κυρίω του φορεί που ασχολούνται με ανθρωπίνα δικαιώματα. Για να έχουν ε, αυτοί οι φορεί δυνατότητα να λειτουργούν πλήρω, ε, θα πρέπει να υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών στην Αφρική. Πρώτη πρόκληση, κυρία Πρόεδρε, τη Αφρικανική Ενώσεω είναι η πρόκληση τη εφαρμογή των μέτρων. Έχουμε άριστα εργαλεία δικαιοδοσία, ε, νομολογία. Έχουμε το Αφρικανικό Δικαστήριο που μπορεί να έχει ποινική αρμοδιότητα και να δικάζει τη διαφθορά, αλλαγή αντισυντεγματική ε, των κυβερνήσεων, πειρατεία κλπ. Η εφαρμογή, η υλοποίηση των μέσων είναι η πρόκληση. Υποφέρει η Αφρικανική Ένωση από χαμηλό ποσοστό εφαρμογής αποφάσεων και συστάσεων. 10% των αποφάσεων εφαρμόζονται. Η κοινωνία των πολιτών. Και ασχολείται μια επιτροπή με αυτό, με την εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτή η επιτροπή επαριθμεί κάποιου λόγου βασικού για τα αίτια, γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσει δηλαδή. Η κοινωνία των πολιτών, όπω σα έλεγα, μπορεί, αν υποστηριχθεί, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να συμμετάσχει στην προσπάθεια την εποπτεία της εφαρμογής των αποφάσεων της Αφρικανικής Ένωσης. Στη βάση πρώτα, σε εθνικό επίπεδο. Τοπικό επίπεδο. Οι χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτές οι χώρες παίρνουν τις αποφάσεις και οι χώρες δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Περί αυτού πρόκειται. η πρόσβαση στα όργανα λήψη απόφαση ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αφρικανική Ένωση δεν έχει εύκολη πρόσβαση κοινωνία των πολιτών σε αυτά τα όργανα. Έχουμε την, Επιτροπή, ε, την Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το δικαστήριο. Η Επιτροπή λοιπόν ωφελήθηκε πολύ από τη συνεισφορά τη κοινωνία των πολιτών. Μέχρι τη δεκαετία των 90 δεν είχε αναλάβει επαρκώς. Είχαμε το 1994 τη γενοκτονία στη Ρουάντα, Φερρυπίν. Πάρα πολλέ παραβιάσει των δικαιωμάτων, πολέμου, συγκρούσει κατά των γυναικών, των παιδιών κλπ. κατά των πληθυσμών. Δεν είχε επιληφθεί η Επιτροπή αυτά τα θέματα, αυτών των θεμάτων. Εδώ και δέκα χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, αυτή η Επιτροπή μετά από μια δεκαετία σήμερα μπαίνει στο θέμα το αυτό των καταγγελιών, καταγγέλει και ελέγχει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε το εξή. Η, η, κοινωνία των πολιτών, η ΜΚΟ, έχουν ένα βήμα τον ΜΚΟ που ετοιμάζει τις συνόδους της Αφρικανικής Επιτροπής του Τοπικών Δικαιωμάτων. Συνεδριάζεται δύο φορές το χρόνο, συμμετέχουν πάνω από 200 μέλη. Είναι κινητήρας καύσιμο για την Επιτροπή, συζητούν τα πάντα. Εκτίθενται οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα σχέδια ψηφισμάτων και συστάσεων συζητούνται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γίνονται πολλέ συνομιλίε. Ετοιμάζονται εναλλακτικέ εκθέσει. Οι ομάδε συμφερόντων προτείνουν θέματα. Οργανώνται παράλληλε εκδηλώσει στο φόρουμ. Η ΜΚΟ που δεν έχουν πολλά χρήματα. Ε, δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να συμμετάσχουν στο, στο φόρουμ γιατί λιγοστεύουν τα μέσα που διαθέτουν. Παρόλα αυτά ε, υπάρχει μεγάλη σημαντική τεκμηρίωση της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να βοηθήσει στου προσπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχουν πρόσβαση στο φόρουμ και να βοηθούν στην προετοιμασία των συνόδων τη Αφρικανική Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και το Αφρικανικό Δικαστήριο. Και εκεί θα έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση εύκολη. Αλλά υπάρχουν εμπόδια για την κοινωνία των πολιτών. Το άρθρο 34.6. Έγιναν 22 έρευνε. Για πολλέ έρευνε υποχρεούται το δικαστήριο να λέει δεν έχει αρμοδιότητα διότι η χώρα δεν έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο. Η χώρα τούτος δεν έκανε την ειδική δήλωση. Υπάρχει αποτελμάτωση σήμερα. Το θέμα της αρμοδιότητας. Λόγω του άρθρου 34.6. Το άρθρο 34.6 ίσως μας οδηγήσει τελικά στο να μην μπορούμε να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Και η γεωγραφική πρόσβαση είναι προβληματική να πάει κανεί ε, σε μακρινέ απόμακρες περιοχέ. Η πρόσβαση οικονομική επίση είναι πρόβλημα για τα θύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να βοηθά τα θύματα ε, να ατυχούν ε, βοήθειας οικονομικής μέσω ταμείου. Ετέθη το θέμα, ήμουν παρόν, στα πλαίσια της προετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου του δικαστηρίου. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους του δικαστηρίου, μέσω του προγράμματος υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης να υποστηρίξει τα θύματα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δικαστήριο. Πρέπει το δικαστήριο να γίνει προσβάσιμο στου πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών, στις γυναίκες, στα παιδιά, στους πληθυσμού, στους ντόπιου. Αυτό είναι το μήνυμα θα πρέπει να δέχεται αιτήματα, υποθέσει από παντού το δικαστήριο, ξεκινώντα από την Αφρικανική Επιτροπή των Λαών και των Δικαιωμάτων Ανθρωπίνων. Δεν μπορούν μόνο οι χώρε να κάνουν δηλώσει. 48 χώρε για τις οποίες, στις οποίες δεν μπορούν οι πολίτες και οι ΜΚΙΟ να προσφύγουν στο δικαστήριο. Έστειλε δύο υποθέσεις στο δικαστήριο η Επιτροπή. Εγώ ε, μία παρέπεμψα. Δύο υποθέσεις δεν είναι πολλές που, που δόθηκαν στο δικαστήριο από την Επιτροπή. Να υπάρχει τέτοιο κενό, τέτοιο χάσμα μεταξύ, έπρεπε να υπάρχει μάλλον διασύνδεση μεταξύ Επιτροπής και Δικαστηρίου καλύτερη, που δεν υπάρχει. Υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Λίγιο χρόνος μου, κυρία Πρόεδρε. Προσπαθώ να συνοψίσω αυτά που λέω υποστήριξη τη Κοινωνία των πολιτών, όπως έλεγα, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία των φορέων των αρμοδίων. Θα πρέπει η Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη ε, πριν να υποβάλει ψήφισμα. Και να διατηρήσει πρέπει να είναι ανεξάρτητη η Επιτροπή. Πρέπει να υπομίζεται τις ευθύνες της. Να υποβάλει τα ψηφίσματά της ανεξάρτητα διότι, αυτό επηρεάζει και την αξιοπιστία του Αφρικανικού συστήματο για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να τεκμηριώνονται όλε οι παραβιάσει των διαπιστωμένων, να, να καταγράφονται οι παραβιάσει που διαπιστώνονται. Θα πρέπει γι' αυτό να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, καταρτιστούν οι διάφοροι φορεί τη κοινωνία των πολιτών. Ε, προγράμματα που είχαν ξεκινήσει έχουν διακοπεί Γινόταν κατάρτιση των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρηματοδότηση έχει διακοπεί και δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάρτιση. Ένα προσπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα φορέα τη κοινωνία των πολιτών, τι μπορεί να κάνει αν δεν έχει κατάρτιση και αν δεν μπορεί να τεκμηριώσει σωστά μία παραβίαση ή δεν μπορεί να ετοιμάσει μία ε, ένα ψήφισμα ή να πάει να μιλήσει στο δικαστήριο. Χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται τεχνική για να παρουσιάσει μια υπόθεση. Χρειάζεται μια βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει του φορεί κοινωνία των πολιτών να καταρτιστούν στη χρήση των περιφερειακών εργαλείων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρήση των διαφόρων εργαλείων και οργάνων που έχει η Αφρικανική Ένωση. Πολλέ φορέ δεν χρησιμοποιούνται παρκώ τα εργαλεία αυτά λόγω έλλειψη γνώση από την κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει το πρόγραμμα ευαισθητοποίηση και αυτοπροώθηση, κάτι που κάνετε, κυρία Κούφο, και το δικαστήριο κάνει και, η προκά... και ο προκάτοχό σα έκανε. Το δικαστήριο όμω πιστεύουμε κινείται. Πήγατε στο Μπουρούντι, σε Νεγάλη, τέσσερι χώρε επισκεφτήκατε. Αυτό δεν αρκεί το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων του δικαστηρίου θα πρέπει να είναι πιο γεμάτο, να πηγαίνετε σε πιο πολλές χώρες και να συναντάτε και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πρόγραμμα μέσω των μέσων ενημέρωσης, μέσω της τεχνολογίας, Twitter κλπ. Να διαδίδετε το μήνυμα, να πείτε θα έρθει το δικαστήριο. Και έτσι η κοινωνία των πολιτών θα μπορεί να προετοιμαστεί για την συνάντηση, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα θέλαμε να σας πούμε, Υπάρχουν πολλά μπορούμε να πάθουμε από το δικαστήριο. Θα πρέπει να ξέρουμε πώς μπορούμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Και κλείνοντα, θα πρέπει να έρθουν τα πολιτικά και νομικά εμπόδια, τα τεχνικά και οικονομικά εμπόδια για την ε, κίνηση των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο είναι δύσκολο να προσφύγει κανείς στη δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρέπει να επιτραψούμε στην ε, Αφρικανική Ένωση έρθει σε επαφή με τις πολίτες, με την κοινωνία των πολιτών, να ενισχυθεί το δυναμικό που έχει η κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση να μπορεί να επιφορτιστεί με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προλάβει τις παραβιάσεις, να προλάβει τα σοβαρότερα εγκλήματα. Χωρί κοινωνία των πολιτών που θα είναι ισχυρή, τα όργανα τη Αφρικανική Ενώση, όπω η Αφρικανική Επιτροπή, όπω το Δικαστήριο, όπω το Οικονομικό Κοινωνικό Συμβούλιο, δεν θα είναι σε θέση να πετύχουν του στόχου του τα δικαιώματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά αλλά και τα πολιτισμικά. Και οι πληθυσμοί της Αφρικής στην τεράστια πλειοψηφία τους δεν θα μπορούν να βγουν από τη φτώχεια. Θα συνεχίσουν να υποφέρουν στη φτώχεια, από την ασθένεια, από την ανεργία για τους νέους, από τους βιασμούς για τις γυναίκες, από τον αποκλεισμό. Η Αφρικανική Ένωση για τις μειονότητες, η Αφρικανική Ένωση αναπτύχθηκε πολύ προηγουμένω, αλλά οι χώρε δεν σέβονται τι αποφάσει αλλά και πολύ λίγες αποφάσεις και συστάσεις εφαρμόζουν. Φανταστείτε ότι κάποιες χώρες δήλωσαν ότι δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις του Αφρικανικού Δικαστηρίου. Δεν δεσμεύονται, αυτό δήλωσαν. Υπάρχουν, δεν σέβονται τα κράτη ούτε τα μέτρα τα, που, δεν, που εμποδίζουν τα μέτρα, τα συντηρητικά μέτρα. Ε, Λοιπόν, έχουν επικυρωθεί τα μέσα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι, πρέπει να βοηθήσει. Είναι τέρος μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας συνδράμει, βοηθά την Αφρικανική Ένωση, πρέπει να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Ε, είναι προς τιμήν σας η οικονομική προσπάθεια που γίνεται, προς το καλό των πληθυσμών μας. Και γι' αυτό χρειάζεται σχέση πιο πολιτικής ε, χρειάς πιο, ε, με την Αφρικανική Ένωση. Το να επερασπίζει τα δικαιώματα κάποιος του αλουνού είναι, σημαίνει αφιέρωση ε, στον άλλον. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε προς τους άλλους, προς τους αφρικανικούς πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ. Χρειάζεται ενίσχυση δικαιοσύνη. για να μην πρέπει να πολεμούν μόνο τους οι πληθυσμοί δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική σας παρέμβαση σε κάποια από τα θέματα που επισημάνατε στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνεισφέρει όπως καταρτίζοντας για την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή με την ε, συνεισφορά της η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θύματα ώστε να υπάρχει ένα ταμείο για την προστασία των θυμάτων. Κάτι παρόμοιο υπάρχει για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Είναι το Εθελοντικό Ταμείο Υποστήριξης Θυμάτων όμως και η εξωτερική υπηρεσία διπλωματικής ε, δράσης ε, μπορεί να μας ε, δώσει περισσότερα στοιχεία πώς μπορεί να υποστηριχθεί αυτό το έργο σε σχέση με την Αφρικανική Ένωση. Έχουμε την κυρία Κορέα ανάμεσά μας να μας τα εξηγήσει αυτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε να παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρατε, πρόσφατα Είχαμε και την ενημέρωση από την υπηρεσία μας ε, για την έκβαση του ε, διαλόγου για τα δικαιώματα του ανθρώπου με την Αφρικανική Ένωση που έγινε το Νοέμβριο 2012 και κάποια από αυτά τα σημεία συζητήθηκαν αυτά τα οποία συζητούμε και εδώ σήμερα. Και είχαμε και άλλες ε, χρήσιμες παρουσίες. Δυστυχώς η υπηρεσία Μπαντζού δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Όμως ελπίζουμε ότι στον 10ο γύρο που θα προετοιμαστεί θα προβλέπεται και θα υπάρχει και η συμμετοχή αυτή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Αφρικανική Ένωση για την θέσμηση, θεσμοθέτηση αυτών των πρωτοβουλειών που ανελήφθησαν. Έχουμε ένα ολόκληρο πλωστάσιο, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Αφρική. Έχουμε επιπρόσθετα μια στρατηγική για τα δικαιώματα του ανθρώπου για την Αφρική. Είδαμε και την χάρτα <clears throat> για τη δημοκρατία, τις εκλογές και τη χρηστή διακυβέρνηση επίσης. Αυτή η στρατηγική, αυτό το πενταετές πρόγραμμα δράσης θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σίγουρα όταν θα έχουμε τη στιγμή να υποπτεύσουμε και να ε, σταθμίσουμε την επίτευξη αποτελεσμάτων σε σχέση και με την στρατηγική που βρίσκεται υπό εξέλιξη. παρόλε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα όργανα της Αφρικανικής Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου για την εκτέλεση της εντολής, Καλοχαιρετίζουμε την Επιτροπή Μπαντζού για τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί σε σχέση με κυβερνήσεις της Αφρικής, για παράδειγμα τη σε σχέση με την κυβέρνηση της Αιθιοπίας. Είναι ενθαρρυντικό και το ότι η Ρουάντα έχει πρόσφατα υπογράψει μια διακήρυξη δίνοντας πρόσβαση στις ΜΚΟ σε τέτοιου είδους δικαστικές υποθέσεις, επιπρόσθετα με τις άλλες είναι θετικό ότι η ε, Αφρικανική Επιτροπή ε, παϊόντων ε, όσον αφορά τα θέματα των παιδιών έχει δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της. Έχει σημειωθεί λοιπόν αρκετή πρόοδος. Παρόλα αυτά, παρόλη αυτή την πρόοδο, και παρόλη την δομή, την αρχιτεκτονική δομή που υπάρχει για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Αφρική, υπάρχουν πολλέ προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν θα υπησέλθω σε όλα αυτά, αλλά λόγω πολιτικ... απουσία πολιτική βούληση από διάφορα αφρικανικά ε, κράτη να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου, με την ομολογία και ακόμα και με την ε, ανεπαρκή στελέχωση από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού παρέχουμε συνδρομή σε αυτά τα όργανα. Ελπίζουμε, ευελπιστούμε ότι αυτή η συνδρομή θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συντονιστική δράση και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Διπλωματικής Υπηρεσίας να συνεχίσει η παροχή αυτής της ε, βοήθειας. Τα επόμενα χρόνια, σε σχέση με την Παναφρικανική αυτή συνιστόσα, αυτό το μέσο θα δώσει τη δυνατότητα να βοηθηθεί η προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχιτεκτονική της Αφρικανικής Ευρωπαϊκής για όλα αυτά. Σημειώνουμε λοιπόν την έκκληση του καθηγητή να υποστηρίξουμε για παράδειγμα το φόρουμ των ΜΚΟ, η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα εκστρατείε ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε με σοβαρό πνεύμα. Έχουμε ευκαιρία να το κάνουμε ούτω ή άλλω και να τα εφαρμόσουμε. Επιπρόσθετα θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε αυτά τα θέματα στα τακτά πλαίσια των διαλόγων που έχουμε με τα κράτη τη Αφρικανική Ένωση. Και ενώ ο διάλογο με την Αφρικανική Ένωση παραμένει η καλύτερη πλατφόρμα για να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτά τα άρθρα, σε αυτά τα θέματα, υπό το άρθρο 8 τους εταίρους μας της Αφρικανικής Ένωσης θα προσπαθήσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα της επικύρωσης του πρωτοκόλου για παράδειγμα για τη χάρτα για την δημιουργία ενός δικαστηρίου ή και για τις δυνατότητες να έχουν πρόσβαση η ΜΚΟ στα τεκτενόμενα. Φυσικά όσον αφορά τα θύματα και όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχουμε το μέσο αυτό για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την προαγωγή αυτών των θεμάτων και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το, να χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Thank um, Σας ευχαριστώ. Θα θέλατε εσείς να παρέμβετε από πλευράς μελών, παρακαλώ. Όχι, κανείς. Έχω μια ερώτηση η οποία δεν συσχετίζεται τόσο στα θέματα επικυρώσεων και εφαρμογής, αλλά περισσότερο θα ήθελα να έχω την δική σας πολιτική άποψη επ' αυτών. Υπογραμμίσατε πόσο σημαντικό είναι βέβαια να καταπολεμηθεί η ατιμορρησία για όλες τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και για τα πολύ σοβαρά εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας. Υποστηρίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δράση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου βέβαια. Και τακτά, σε τακτά διαστήματα στις συζητήσεις ακούμε από εκπροσώπους, κυρίως εκπροσώπους κυβερνήσεων τα σχετικά από την Αφρική, ότι είναι προκατηλημένο, λένε, ομά κιόλα αυτό το δικαστήριο. Εξετάζει μόνο περιπτώσεις κατά πρώην στρατιωτικών ε, κυβερνήσεων στρατιωτικής διοίκησης αφρικανικών χωρών. Ξεχνώντας ότι υπάρχουν και αφρικανικές χώρες οι οποίες προσφεύγουν στο δικαστήριο και ζητούν τη σύνδρομή του. Τώρα, ακολουθώντας αυτό, βλέπετε να υπάρχει μια συνέχιση αυτή της επανάληψης ε, σε σχέση με μια προκατηλημένη ας το πω έτσι τοποθέτηση ή υπάρχει εδώ διαφορετική αξιολόγηση του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο αυθεντικό έργο που επιτελεί ε, συνδράμοντας ε, για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη και την τιμωρία όχι μόνο κάποιων αλλά όλων των υπεύθυνων. Ευχαριστώ. 13 2012 το Δεκέμβριο του 2012 οργανώθηκε στην Αφρικανική Ένωση κατόπιν αιτήματο συγκεκριμένων πρέσβεων ένα σεμινάριο για την διεθνή ποινική δικαιοσύνη και συμπεριλαμβάνονταν στους συμμετέχοντες πολλές χώρες, καμιά εικοσαριά χώρες. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια ακρόαση για το ίδιο θέμα, για τη δικαιοσύνη και πάλι. Και τα περισσότερα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης συμμετείχαν Δηλαδή, το λέω αυτό για να σας πω ότι μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Και όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν κράτη που ε, προσέφηγαν ε, στο ποινικό δικαστήριο. Αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση μεταξύ των Αφρικανικών κρατών και του ποινικού δικαστηρίου. Σε αυτό το σεμινάριο πολλοί πρέσβεις είπαν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν θέλησε να ανταποκριθεί σε ένα αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Ρώμης και αυτό κάπως ε, έθεσε φραγμού στη συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τη ε, Αφρικανική Ένωση και η πολιτική διώξεων του προηγουμένου εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ίσως ε, ήταν τέτοια που έδινε μια εικόνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου διαφορετική, ότι είναι η δικαιοσύνη των Λευκών έναντι των Αφρικανών. Δόθηκε μια τέτοια εικόνα. Ε, σήμερα Ε, ξεχνώ το όνομά ε, αλλά η εισαγγελέα που είναι υπεύθυνη ε, είναι μια γυναίκα από την Αφρική που είναι σημαντικό πρόσωπο και είναι σημαντικό να είναι ένα διεθνές το δικαστήριο, το ποινικό δικαστήριο που να ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα και στις περισσότερες περιπτώσεις κράτη ζήτησαν από το ποινικό δικαστήριο στην περίπτωση του, της ακτής του ελεφαντοστού, του κ. Μπαμπά κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι αυτό το δικαστήριο διώκει μόνο Αφρικανούς και πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο. Πάντως είναι και αυτό ένα θέμα που μας απασχολεί. Η συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση είναι σημαντική θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Αφρικανική Ένωση και αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα που θα επιτρέψει καλύτερο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης. Και θα πρέπει τα κράτη της Αφρικής να εκδικάζουν τις υποθέσεις στη χώρα τους με σωστό τρόπο για να αποφεύγουν την προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά τα δικαστήρια επιτόπου για να διώκονται τα εγκλήματα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Αυτά ως απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται καταρχήν τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης εφόσον λειτουργούν και μόνο αν δεν λειτουργούν τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης τότε θα παρέμβει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και είναι κρίμα διότι μέχρι πριν από πέντε χρόνια το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θυμάμαι ήταν το 2010 στην Καμπάλα υπήρχαν κάποια ε, σχέδια να ανοίξει ένα περιφερειακό γραφείο στην Αντίσα Μπέμπα για να βελτιωθεί το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Χθε, όταν ο Δ. Λαμίνη Τσούμα, πρόεδρος ε, της Επιτροπής Αφρικανική Ένωση, είπε ότι οι προκλήσει τώρα ε, θα πρέπει να τεθούν στον ορίζοντα του 2050, σκέφτηκα ότι ίσως και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να είναι μια σκέψη αυτή, δηλαδή κάπως η δομή του δικαστηρίου να περιλαμβάνει κάποια σχέδια ανάπτυξης και στην Αφρική. Τώρα, μιας και είστε εδώ παρόν για να υποφεληθούμε, θα ήθελα να πω το εξή. Αποφασίσαμε ε, στην Επιτροπή μα να ασχοληθούμε με μία έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλέον επίγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο ΣΑΧΕΛ από την κοινωνία των πολιτών όπως τη γνωρίζετε εσείς. Εμείς συζητήσαμε την κατάσταση και στο Μάλι και στις γειτονικές χώρες και είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Και μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο συνάδελφος κύριος Ρώτα επίσης θέλει να κάνει μια ερώτηση. Θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απελευθερώθηκαν οι Γάλλοι ε, όμοιροι, να σας πω αυτά τα νέα, είναι ικανοποίηση. Και ήθελα να το πω αυτό στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό να σας θέσω μια ερώτηση. Μιλάμε για το Σαχέλ. Θα ετοιμάσουμε την έκθεση, θα είναι έξοχη η έκθεση. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς το Σαχέλ. Η θέση των Σαχέλ είναι στην υποσαχάρια ζώνη. Πόση απόσταση, πόσες χώρες. Ετοιμάζουμε έκθεση και δεν ξέρουμε πόσες χώρες αφορά το Σαχέλ. Α, πάει από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό. 13 χώρες θα είναι αυτή η περίπτωση. Για να γίνει μια έκθεση πρέπει να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και για ποιες ε, χώρες ε, μιλάμε. Νομίζω ότι ο ορισμός γεωγραφικός του Σαχέλ είναι τα όρια της Σαχάρας. Πολιτικά σήμερα, γεωπολιτικά, το Σαχέλ ξεπερνά τα όρια κατά πολύ της Σαχάρας. Το Καμερούν σήμερα και μας δώσατε και πολύ καλά νέα, κυρίως για την απελευθέρωση, κυρίως των παιδιών. Τέσσερα παιδιά. Ένα είναι πέντε ετών, το άλλο δώδεκα που απελευθερώθηκαν. Και αυτό μας κάνει καλό στην καρδιά, όμως δεν λύνει το πρόβλημα του Σαχέλ. Πάει από τον ωκεανό μέχρι τη Σομαλία και την Κένια. Είναι η Αφρική υπό Σαχάρια. Δεν είναι μόνο το Σαχέλ, είναι η Αφρική. Περί της Αφρικής πρόκειται. Το Καμερούν, είναι στην Κεντρική Αφρική το Καμερούν. Και αυτό πλήττεται. Πλήρως. Είναι σημαντικό η έκθεση να, είναι, να έχει το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο και υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Είναι πολύ αδύναμες οι χώρες Αν πάτε και να δείτε τον, τον κατάλογο με την ε, ανάπτυξη, οι φτωχότερες χώρες στον κόσμο θα δείτε ότι είναι στο Σαχέλ. Οι πιο φτωχές χώρες είναι σε αυτή τη ζώνη του Σαχέλ. Εδώ και 20 χρόνια το Σαχέλ είχε πληγεί πολύ άσχημα από την ξηρασία. Και είναι ανύπαρκτη σχεδόν η γεωργία σε πολλές χώρες, διότι προχωράει έρημος και με μεγάλα βήματα. Και βέβαια αυτό συνδέεται και με τα προβλήματα τα κλιματολογικά. Εγώ είμαι Σενεγαλέζος, ε, είμαι από το Σαχέλ. Το Σαν Λουί, στη Σενεγάλη, πόλη μου, είναι έρημος. Έχουμε την έρημο στη Σενεγάλη τώρα. Η μισή Σενεγάλη είναι έρημος. Και αυτή η πρόοδος, η γεωγραφική της ερήμου είναι παράγον πολύ σημαντικός φτώχειας. Ε, για χώρες που έχουν μπει σε προγράμματα διαθροτικής προσαρμογής ε, και στο Μάλι και λοιπά. Λοιπόν, και έχουν γίνει πάρα πολλές περικοπές οικονομικές λόγω πολιτικών ε, προσαρμογής και οι πληθυσμοί έχουν υποφέρει από τις διάφορες προσαρμογές. Η παιδεία έχει υποφέρει, η υγεία έχουν πληγεί όλοι αυτοί οι τομείς. Και σήμερα ναι, έχουμε και τα προβλήματα όλων αυτών. Τα συστήματα αμήνη δεν μπορούν να δράσουν, ο στρατό έχει πληγεί, φτώχεια που η φτώχεια γεννά είναι γόνιμο έδαφος για κάθε είδους πρόβλημα. Λένε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν πάνω από 100.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι. Ε, διάφορα πτυχία και υψηλού επίπεδου πτυχία κοινά ανεργία. Το πρόβλημα είναι καταρχάς οικονομικό, πριν να είναι πρόβλημα άμυνας, Δεν μπορούμε να βάλουμε ευρωπαϊκό ή γαλλικό στρατό σε όλο το Σαχέλ. Αυτό είναι αδύνατο. Η μισή Αφρικανική Ήπειρος θα πετούσε 13 χώρες. Καμία κοσαριά χώρε θα έπρεπε να καλύπτονται έτσι. Δεν μπορούμε να στέλνουμε παντού τεύματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η ρίζα του κακού, τα οικονομικά προβλήματα. Η νέα, οι νέοι, συγγνώμη, τι θα προτείνουμε στου νέου. Δεν προτείνουμε πολλά. Δεν έχουν πολλέ ελπίδε οι νέοι. Δεν είναι ευρύ ορίζοντα για του νέου. Οι γυναίκε. Διότι έχει ε, πρόσωπο γυναίκα στη φτώχεια, κυρίω εκεί. Η πρόσβαση των γυναικών στη γη είναι δύσκολη. Η δημογραφική η έκρηξη είναι πρόβλημα. Η προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια ε, είναι πολύ περιορισμένη. Χρειάζεται πιο ολιστική, σφαιρική προσέγγιση να λάβει υπόψη πολλούς παράγοντες, τους οικονομικούς παράγοντες, τα αίτια τα οικονομικά. Σήμερα βλέπουμε τα αίτια. Κακή διακυβέρνηση, ε, χρόνια διαφοράς ενδημικής επίσης είναι αίτια, όπου είναι πολύ λίγα τα χρήματα και οι περισσότεροι δεν έχουν καν τα ελάχιστα εισοδήματα, τα ελάχιστα χρήματα που απαιτούνται για να ζήσουν, τα μέσα για να ζήσουν. Λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα έχουν στη διάθεσή τους. 50 λεπτά ε, Λοιπόν, κάτω από 300 φράγκα κεντρικής Αφρικής. Οι γυναίκες, οι μητέρες οικογενειών δεν μπορούν να θρέψουν τα παιδιά τους, τα μωρά τους. Αυτό είναι. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Thank you. And now we are coming to... Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνεται εδώ αυτός ο γύρος αυτής της συνεδρίασης. Θα ήθελα να ζητήσω από τη δικαστήνα, να πω στη δικαστήνα στην Αρούσα να σας ευχαριστήσουμε που παραμείνατε κοντά μας. Αν έχετε κάτι που θα θέλατε να μας πείτε στο τέλος. Um, two, two issues. Um, the first one, I just needed to clarify something and concerning the relationship between the court and the Banjul Commission, which um, I always wonder why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 the, European Parliament. thank you and uh, thank you also from our side that you could... Σας ευχαριστούμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που λάβατε μέρος σε αυτή την ακρόαση. Είτε και ελπίζω να σας ξαναδούμε στο μέλλον, ε, είτε παρούσε εδώ, είτε μέσω βίντεο διάσκεψης και πάλι. Ευχαριστούμε και τον καθηγητή Φάλ και θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μούσνιξ, Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είχε πάει στην Ελλάδα αυτός. συζητήσαμε τα θέματα της περιοχής ΑΣΕΑΝ, ακούσατε και ένα τμήμα της ακρόασης που κάναμε για την Αφρικανική Ένωση και τώρα έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης και δεν είναι πρώτη φορά που ενημερωνόμαστε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και που προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας για να μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δικά σας ευρήματα και τις δικές σας συστάσεις για να ενισχύσουμε τη δική μας δουλειά. Έχουμε κάνει συνεδριάσεις και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και κάναμε και μια συνάντηση πριν από ένα χρόνο περίπου Μα είχατε πει ότι θα προτιμούσατε να αφήσουμε να περάσει λίγο χρόνο για να έρθετε, στην Επιτροπή μα, γιατί αναλάβατε καθήκοντα πριν από ένα χρόνο και θέλετε να, έχετε διαμορφώσει κάπως τη θέση σας για να ξέρετε τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε. Και μάλιστα, επί τη ευκαιρία θέλω να πω ότι ενημερώσατε και την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο Βερολίνο, στη χώρα μου, για σχετικά θέματα σε μια επίσκεψή σας ε, την οποία έρχεστε και πριν ε, να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική σε άλλους, καλό θα είναι να βάλουμε τάξη στη δική μας χώρα κάθε φορά, γιατί και εκεί ξέρω ότι υπάρχει μία δεσμευτική μειοψηφία σε σχέση με τα θέματα προτεραιότητά σας. Η Επιτροπή μας, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως πολλά θέματα τα οποία μπορούμε να συζητάμε και ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μας επισκέπτεται και χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε ε, μια αποστολή στη ΦΥΡΟΜ και θα γίνει και μια αποστολή στη Σερβία φέτος. και μιλάμε για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στι γειτονικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητάμε και με του διαμεσολαβητέ από τι γειτονικέ χώρε. Σα δίνω το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη μου ε, παρέμβαση εδώ στην Επιτροπή, ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου πέρυσι τον Απρίλιο και ε, ιδίω όταν είστε στο Στρασβούργο ευχαρίστω να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα σα. Θα μπορούσα να σα πω δύο λόγια και για το δικό μου το έργο και για τι προτεραιότητε που έχω εντοπίσει και που έχω αρχίσει να παρακολουθώ. Το γραφείο μου είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, αμερόληπτος, που ε, βοηθά τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης να πληρούν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν λέω ανεξάρτητος θεσμός σημαίνει ότι δεν παίρνω οδηγίες ούτε από χώρες, ούτε από Γενικό Γραμματέα, ούτε από, από την κοινοβουλευτική συνέλευση και όταν λέω αμερόληπτη αρχή σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθώ και με τα 47 κράτη-μέλη, πράγμα που είναι μια πρόκληση και παράλληλα είναι και τιμή για μένα, διότι πολλοί κατηγορούν τα θεσμικά όργανα ότι κρίνουν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ πρέπει να εξετάζω όλες τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης για να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, έχω φοιτεία εξαετή, επομένως έχω καλύψει ένα από τα έξι χρόνια της θητείας μου αυτό το οποίο κάνω είναι ότι πηγαίνω σε κάποιες χώρες, εντοπίζουμε κάποια θέματα προτεραιότητας, συναντάμε την κοινωνία των πολιτών, υπουργού, διαμεσολαβητές, μέλη του Κοινοβουλίου και συντάσσουμε μια έκθεση με τις συστάσεις μας και στη συνέχεια παρακολουθούμε την κατάσταση. Συνεχίζω να έχω επαφές με υπουργούς, ε, κάνω και νέες επισκέψεις στη χώρα, συναντώ βουλευτές, ε, μιλώ με τα μέσα ενημέρωσης και τα κριτήρια για την επιλογή μιας χώρας ε, ποικίλουν. Η γεωγραφική ισορροπία είναι ένα θέμα γιατί προσπαθώ να καλύπτω όλες τις περιοχές ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης κάθε χρόνο. Δεν πηγαίνω μόνο στο Νότο ή μόνο στις ανατολικές χώρες. Από ναι, το δεύτερο κριτήριο είναι το πόσος χρόνος έχει περάσει από την προηγούμενη επίσκεψη και το τρίτο κριτήριο είναι το αν υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση που απαιτεί να της δοθεί προτεραιότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά που κάνουμε, πολύ απαιτητική, με πολλές προκλήσεις. Βεβαίως και μπορούμε να συζητήσουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει πολλέ ε, συναντήσει με επιτρόπους Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα θα συναντήσω την Επίτροπο Κρού. Ε, έχω συναντήσει και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και τον κύριο Λαμπρινίδη και θα τον ξανασυναντήσω και σήμερα λίγο αργότερα. Και έχουμε συνεργασία και επιτόπου. Δηλαδή όταν επισκεπτόμαστε μια χώρα προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να ανταλλάξουμε απόψει για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συμπληρωματικά στοιχεία. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ ε, στενή επικοινωνία για να υποφεληθούμε από αυτή την συμπληρωματικότητα. Θα σα πω ποιε είναι οι μεσοπρόθεσμε προτεραιότητέ μα. Πριν εκλεγώ ω Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τα... Δεσμεύτηκα ότι θα κάνω ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ένα θεσμό που δεν πρέπει να καταρρεύσει υπό το βάρο τη επιτυχία του γιατί θα αρχίσει να διαλύεται ολόκληρο το σύστημα. Και πώς μπορώ να τους βοηθήσω. Καταρχήν πηγαίνοντας σε χώρες που στέλνουν πολλές υποθέσεις στο δικαστήριο. Χώρες από τις οποίες δημιουργούνται κατ' επανάληψη υποθέσεις που φτάνουν στο δικαστήριο. Μερικές φορές υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις, προβληματικές. Παραδείγματος χάρη μία από τις πρώτες υποθέσεις ήταν στην Ιταλία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα σας ενδιαφέρει, αλλά ήταν ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα που αφορούσε τι τις εκλογικές διαδικασίες. Άλλα παραδείγματα η Ρωσία, η Τουρκία, στις οποίες επανέρχομαι αυτή τη χρονιά για να εξετάσουμε την απονομή δικαιοσύνη. Και φέτος ε, για τη Ρωσία και για την ε, Τουρκία θα κάνουμε τέσσερις επισκέψεις και θα γράψουμε τις σχετικές εκθέσεις για την απονομή δικαιοσύνης στη Ρωσία και στην Τουρκία Όσον αφορά τι αποφάσει του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρακολουθούμε υποθέσεις, ε, επισκεπτόμαστε τις χώρες, μερικέ φορέ στην επέτειο ιστορικών αποφάσεων του Δικαστηρίου, ερχόμαστε σε επαφή με υπουργού που πρέπει να εφαρμόσουν κάποιε αποφάσει. Άλλε φορέ ε, δουλεύουμε με τα μέσα ενημέρωση για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τη δουλειά που πρέπει να γίνει και είναι μια συνεχής πρόκληση η δουλειά μας. Ε, είναι ένα συνεχές έργο και ασχολούμεθα με χώρε και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε του Συμβουλίου τη Ευρώπη γενικότερα. Όσον αφορά την δικαστική εξουσία, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά την οικονομική κρίση, η δικαιοσύνη και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη συγκεκριμένα ε, θίγεται κατά πολύ και όσον αφορά τα ένδικα μέσα και όσον αφορά την πρόσβαση ε, σε νομικά μέσα και στους θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει και στην Αλβανία και στη Γεωργία. Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας είναι ένα θέμα προς ε, συζήτηση ε, επί πολλά χρόνια. Θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και στο μέλλον και θα επηρεάσει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθενται προκλήσεις όχι μόνο για το κεκτημένο για τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στην Ευρώπη, αλλά και για πολλά πολιτικά και για πολλά πολιτικά δικαιώματα, ε, περικοπές του προϋπολογισμού ε, και για το σοφρονιστικό σύστημα, είτε υπάρχουν ε, ε, μακρύ χρόνη παραμονής ε, των φυλακισμένων ε, στη φυλακή. Γίνονται προσπάθειες για την αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών που και αυτές θα απαιτούν πόρους και πλήττονται από την περικοπή των πόρων. Έχουμε κάνει πολλές επισκέψεις, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα περιοχές όπου τα μέτρα λιτότητας πλήττουν ε, πολλούς τομείς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Από τις ευάλωτες ομάδες που πλήττονται περισσότερο είναι η Ρώμα. Οι προτεραιότητες τις οποίες εντοπίζουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρωμά είναι οι εξής. Καταρχήν, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του διαχωρισμού της εκπαίδευσης, ε, του ότι τους ε, δίνεται ε, χωριστή εκπαίδευση. Ακόμη ένα άλλο πρόβλημα είναι το καθεστώς του απάτριδος για τους Ρωμά. Αυτό δεν ισχύει μόνο σε χώρες της πρώην Ιουκοσλαβίας, αλλά και σε άλλες χώρες, και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη στάση κατά των Ρωμά και εδώ έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα της καταπολέμησης αυτού της της ε, αρνητικής μεταχείρισης. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε λοιπόν αυτά τα αρνητικά, αυτές τις αρνητικές προκαταλήψεις κατά τον ε, Ρωμά. Ένα άλλο θέμα είναι η μετανάστευση των ε, Ρωμά, κάτι που αφορά πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το θέμα των Ρωμά Υπάρχει πεδίο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γραφείου μου και του Συμβουλίου της Ευρώπης γενικότερα. Χρησιμοποιούμε στοιχεία ε, για τις ευρωπαϊκές χώρες από τους αρμόδιους φορείς και υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα και από ε, το Πρόγραμμα Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών για τις μη ευρωπαϊκές χώρες. Όπως σας είπα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι και η Επιτροπή έχει μιλήσει για στρατηγικέ ενσωμάτωση των Ρωμά και θα θέλαμε να δούμε περισσότερε πολιτικέ για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Επίση, ε, θα ήταν θετικό να εφαρμόζεται η οδηγία, καλύτερα η οδηγία ε, για την ισότη, τη φιλετική ισότητα. Μία από τι χώρε που έχουμε στην έκθεσή μα και που μπορεί να σα ενδιαφέρει ε, του προσεχεί μήνε είναι η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Υπάρχουν πολλά θέματα τη χωριστή εκπαίδευση για του Ρώμα ε, προσπάθειες ε, για περιορισμό ε, των Ρωμά ώστε να μην φεύγουν από τη Φιρόμ και πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζητούν άσυλο. Σε πολλές περιπτώσεις δημεύονται, τα, τα, τα διαβατήριά τους από τις αρχές Μερικές φορές ε, μιλάμε για διευκόλυνση της ε, πολιτικής χορήγησης βεβαιώσεων ε, διαβατηρίου, αλλά γίνεται με προβληματικό τρόπο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση των Ρωμά λοιπόν είναι προβληματική. Πολλές φορέ και στη χώρα προέλευσή τους και σε άλλες χώρες υπάρχουν απαγορεύσεις εξόδου, υπάρχουν υποχρεωτικές επιστροφές και το θέμα της κατάσταση των διαβατηρίων τους ε, είναι πραγματικά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε μόνο στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας, αλλά και στη Σερβία και στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη. Ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό είναι η προστασία των μέσων ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένης και της ε, προστασίας των δημοσιογράφων. Εδώ ασχολούμαστε και με τις τεχνολογίες και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα όπου αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους ζητήματα. Πήγαμε μαζί με την Τούνια Μιάτεβιτς ε, ε, σε ένα φόρουμ ε, για την ελευθερία των μέσων. Επισκεφθήκαμε φυλακισμένους στο Αζερβαϊτζάν και μαζί με την Επίτροπο Κρούζ συζητήσαμε με δημοσιογράφους από το Αζερβαϊτζάν για την ελευθερία έκφρασης. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας γιατί από κοινού αυτά τα οποία είπαμε είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι αν τα λέγαμε χωριστά ο καθένα. Και στο Αζερβαϊτζάν θα επανέλθουμε για μια πλήρη έκθεση για την ε, ελευθερία έκφραση και για την ελευθερία του συνέρχεστε. Κλείνοντα, θα ήθελα ε, να τονίσω ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι εθνικές δομές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για μας είναι σημαντικοί εταίροι. Όσον αφορά τη δική μου θητεία ε, συχνά οργανώνουμε ε, συζητήσεις ε, με τους υπερασπιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων. Τους συναντάμε και στο Στρασβούργο όταν έρχονται για την κοινοβουλευτική συνέλευση και σε, σε επισκέψεις που κάνουμε στις διάφορες χώρες. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία τους, αξιολογούμε τις απειλές ή τις επιθέσεις εναντίον τους. Ε, και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Όπω επίση και οι εθνικέ δομέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική εταίροι για μα, γιατί του θεωρούμε σημαντική πηγή πληροφοριών και είναι φορεί που μπορούν να προωθήσουν την, ε, τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα. Έχουμε τακτικέ επαφέ μαζί του και στο Στρασβούργο και σε αποστολέ μα στι διάφορε χώρε και προσπαθούμε ε, να συνεργαζόμεθα με, τις, ε, με τους διάφορους ε, φορείς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη δική μας συνάντηση θα συναντηθώ και με τον διαμεσολαβητή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Μιας και συζητάμε τα θέματα συνεργασίας. Να σας πω τις χώρες που θα επισκεφθούμε τους επόμενους μήνες. Δεν έχουμε επισκεφθεί ακόμη την Μολδαβία. Θα πάω και στην υπερδνηστερία. Αζερβαϊτζάν, Ρωσία, Τουρκία, Γεωργία. Θα επισκεφθώ επίσης και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εστονία, Ισπανία, και κάποιε άλλε που ακόμη δεν έχουμε ενημερώσει τους πρέσβει τους, επομένως δεν θα το ανακοινώσω τώρα για να το ανακαλύψουν από μια ακρόαση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν αυτές τις χώρες λεπτομερέστερα. Αλλά α περιμένουμε να ακούσουμε τι δικέ σα ερωτήσει πριν απαντήσω. Σε ευχαριστούμε. Υπάρχουν κάποιε ερωτήσει. Έχω και εγώ κάποια ερώτηση. Εσείς παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγεται, λέγοντας πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, να υπάρχει αμεροληψία, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα ήθελα να γνωρίζω επακριβώς από τη στιγμή που διαπιστώνεται το μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα, ποιε είναι οι κυρώσει, όχι μόνο να επισημαίνονται αυτά, αυτό το κάνουμε και εμεί εδώ. Θα ήθελα να ξέρω ποιε κυρώσει επιβάλλεται οι αναβάλουμε για αύριο αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα. Ε, για το ρατσισμό, μιλήσατε για το έργα, την εργασία των παιδιών, ε, αναφέρατε κάποιες χώρες, δεν τις αναφέρατε, τις κατονομάσατε, τις ξέρετε όπως και εγώ, καμιά φορά ε, κατονομάζονται και δεν υπάρχει όμως κύρωση. Δεν είμαι ο Ζωρό και ο Νταρτανιάν που φτιάνει με το σπαθί του για να λύσει τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι χώρες. Η εντολή μου είναι να βοηθώ τις χώρες τα κράτη-μέλη μέσω διαλόγου για να γίνεται μια ανάλυση βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τα, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καμιά φορά έχουμε προγράμματα βοηθείας. Παραδείγματο χάρη αν μια χώρα χρειάζεται κατάρτιση των δικαστών, ε, των εισαγγελέων, μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Η δεμή όλα εξαρτώνται από την καλή βούληση των ε, κρατών μελών δεν είναι στόχος μου, τακτική μου, να επικρίνω για την επίκριση. Θέλω να δείχνω το δρόμο μέσω ανάλυσης βάσει προτύπων προδιαγραφών και αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καμιά φορά μπορούμε να έχουμε επιρροή, καμιά φορά δεν την έχουμε εξαρτάται από το εθνικό πολιτικό πλαίσιο, εξαρτάται από το ενεργασία μας, αν μπορούμε να βρούμε καλό εταίρο, βουλευτή, διαμεσολαβητή, υπουργό, που θέλει να βρει καλύτερη επιχειρηματολογία για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Καμιά φορά η παρουσία μας μπορεί να βοηθήσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν, διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, μία επίσκεψη στη φυλακή απλώς ε, μπορεί να βοηθήσει. Αλλά καμιά φορά είναι και θέμα ευαισθητοποίησης, όχι μόνο των πολιτικών αλλά και του κοινού. Λόγω όλων αυτών όλη η δουλειά μας είναι διαφανής, εργάζομαι πολύ με τα ΜΜΕ και προσπαθώ να επικεντρώσω την προσοχή επί του προβλήματος και πώς πρέπει να γίνει ο χειρισμός του ζητήματος. Αλλά οι κυρώσεις μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, έχει δικαίωμα επιβολής κυρώσεων. Μπορεί να απαιτήσει από ένα κάτω μέρος να πληρώσει αποζημίωση ή να αλλάξει τον νόμο για να αποφευχθούν ε, παραβιάσεις στο μέλλον. Εργαζόμαστε πολύ με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διότι είναι το νομικό πλαίσιο των εργασιών μας αυτό. Και είναι πολύ καλό αυτό για μας, διότι μπορώ να πω στα κράτη-μέλη αυτά είναι τα πρότυπα που δεχτήκατε, νομικές προδιαγραφές, δεν είναι πολιτικές συστάσεις, είναι ε, προδιαγραφές ε, δικές σας και όχι κάποιο οργανισμού του εξωτερικού στον οποίο δεν ανήκετε. several Αρκετά ερωτήματα για αυτά που είπατε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θυμούμε ότι εγκρίναμε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη συνάντηση στο Brighton και είμαστε υποστηρικτικοί στο να ενδυναμωθεί το έργο του δικαστηρίου. Κάποιες από τις αποφάσεις από την ομολογία του ΔΕΚ είναι σημαντικές για το να ενισχυθεί το έργο όπως η ε, απόφαση, η νομολογία σε σχέση με την προσφυγή όσον αφορά την Ιταλία για την, ε, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στην εντολή μας πεθαίνουν άνθρωποι επειδή αποκρούεται είσοδο είσοδος τους, ε, ε, τους αρνούνται είσοδο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εδώ σε σχέση με, την, με το 10 το ίδιο συμβαίνει και στις ανοιχτές θάλασσες. Μπορεί να ζητούν άσυλο και θα πρέπει να βοηθούνται αυτά τα άτομα. Αυτό υποστήριξε πάρα πολύ την πολιτική συζήτηση σε τεράστιο βαθμό αυτή η νομολογία. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει εκθέσεις έχει εκπονήσει εκθέσεις η κυρία Σκίνη και, σωστά προφέρω το όνομα τεκμηρίωσε όταν είχαμε άτομα από τη Λιβύη που αποβίωσαν προσπαθώντας να ε, ε, προσέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν και δεν βοήθησαν ε, και τα σκάφη του ΝΑΤΟ. Το θυμούμε πολύ καλά αυτό. Και όλο το θέμα των μεθοριακών ελέγχων και της υπηρεσίας Frontex να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Καταβάλουμε προσπάθειες για να πετύχουμε αυτό το στόχο στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπατε, αναφέρατε δύο χώρες για τις επισκέψεις σας στη Ρωσία και στην Τουρκία. Έχουμε και μια αντιπροσωπεία που πήγε το Δεκέμβριο στην Τουρκία και πήγαμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι εκπληκτικό πόσες προσπάθειες καταβάλλονται ώστε να μειωθούν αυτές οι περιπτώσεις, να αντιμετωπιστεί ο τεράστιος αριθμός, πόσες προσπάθειες καταβάλλονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο δικαστικό σύστημα εκεί. Εντυπωσιακό αυτό. Επίσης βλέπετε όταν πηγαίνετε εκεί αλλά και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε ένα διαφορετικό επίπεδο όπου αναμειγνύεται το πολιτικό επίπεδο. Οι πολιτικοί ε, ε, παρεμβαίνουν, πράγμα το οποίο ε, αντιβαίνει εντελώς απόλυτα τις ε, άλλες εξελίξεις στην Τουρκία και στην ετήσια έκθεση για την Τουρκία αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η τουρκική πλευρά είναι να ανοίξει αυτό το δικαστικό πακέτο μέτρων, αυτή η δέσμη μέτρων θα το έχουμε και ω θέμα στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή αλλά και στην αντιπροσωπεία μας με την Τουρκία. Θα είναι κύριο ζήτημα αυτό διότι έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για μας. Για την Ρωσία είχαμε και εχθές συζήτηση σχετικά εδώ και με τον ειδικό εκπρόσωπο του ε, Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και τον ειδικό εντεταλμένο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι πιο δύσκολα εκεί τα πράγματα, διότι σε σχέση με τη συζήτηση το τι γίνεται σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ ξεχνάμε να συζητήσουμε κάποιες άλλες πτυχές. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την πτυχή και να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτά τα θέματα. Και από την άλλη πλευρά τα θέματα των τσιγκάνων, των Ρωμά που στην ακρόαση για τη Ρωσία. Καλέσαμε τις ΜΚΟ και συνήθως έχουμε μια ε, μόνιμη ημερήσια διάταξη για τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και συναφή θέματα. Είχαμε δύο προσώπους από την οργάνωση Memorial που μας ε, ε, παρουσίασαν την, κατάσταση των φτωχών και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τόσες διακρίσεις και αποκλεισμού στην Ρωσία. Και επίσης για την κοινότητα των Ρωμάτων Τσιγκάνων που την ίδια αντιμετώπιση έχουν εκεί και για τους Τσιγκάνους ε, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, μια και όλα αυτά δεν είναι δεσμευτικά, να απαιτηθεί από τις κυβερνήσεις να πάρουν αυτά τα κονδύλια και να κάνουν δεσμευτικά κάτι. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται υπό εξέλιξη ούτως ή άλλως ε, ως ε, ζήτημα από πλευράς μας που θέλουμε να ευδοκιμήσει. Και αυτό που είπατε για την κατάσχεση διαβατηρίων ταξιδιωτικών εγγράφων για ανθρώπου που κατάφεραν να φτάσουν σε κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάσχονται μετά τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, τα διαβατήρια. Θα συνιστούσα να ε, δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα ούτω ή άλλω ε, και να το δούμε σε βάθο. Είχαμε και μια ε, προετοιμασία για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων για την αντιπροσωπεία σε σχέση με την αποστολή στην Μακεδονία. Θα έπρεπε αυτού του είδου πληροφορίε να μπορούν να διαχέονται σε σχέση με αυτό το θέμα για την εντολή. Ρώτησε τώρα για τις κυρώσεις ε, ε, προηγούμενα ε, κάποιος και επανέρχομαι στη Ρωσία διότι η σύστασή μας ήταν αυτή σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο γιατί δεν επιβάλλουν τα κράτη-μέλη κυρώσεις ιδιαίτερα στην περίπτωση Μαγνίτσκι βλέπουμε ότι είναι ένας στενός κύκλος ατόμων που είναι υπεύθυνα αυτά τα άτομα για αυτή την κατάσταση και σε σχέση με την κατάσταση του Μαγνίσκη δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι ως Ευρωβουλευτές όταν έχουμε επαφή με κράτη-μέλη. Πώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και τι γίνεται. Όταν διατυπώνουμε τέτοια ερωτήματα δεν δίνονται απαντήσεις, βλέπετε. Επίσης το θέμα των κυρώσεων είναι πολύ ακαθόδες, πολύ ευαίσθητο ε, και δυσχερές ε, πολιτικά. Ε, πώς μπορεί να προχωρήσει κανείς. Αν υπάρχουν όμως στοχοθετημένες κυρώσεις, ίσως αυτό μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Κίνκα παρακαλώ. Sorry, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπούμε που καθυστέρησα έπρεπε να συμμετάσχω σε κάποιες ψηφοφορίες σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω εξ ολοκλήρου την παρουσίαση. Έχω μια ερώτηση όμως. Οι ε, εθνικές ε, γλωσσικές ε, μειονότητες στην Ευρώπη παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τι γίνεται, τι τεκταίνεται στο Συμβουλίο της Ευρώπης και έχουν μεγάλη σπουδαιότητα αυτά τα θέματα, τα γλωσσικά, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι υπάρχει ελπίδα θα υπάρξει επίλυση των προβλημάτων τους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ερώτησή μου συγκεκριμένα, αν υπάρχουν τέτοιου είδους εξειδικευμένα ειδικά προβλήματα, και αν όλα δεν είναι τόσο τέλεια. Έχουμε βέβαια τα γενικά πλαίσια, αν όμως υπάρχουν και όταν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που αναφύονται, τι μπορεί συγκεκριμένα να γίνει και πώς μπορεί κάποιο θέμα να προχωρήσει. Σας ερωτώ, έχετε την πρόθεση να επικεντρωθείτε και σε αυτά τα θέματα γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη και τι συγκεκριμένα εξειδικευμένα πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και μπορείτε να κάνετε εσείς θα δώσω απάντηση σε αυτά που θέσατε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Μετανάστευση. Συμφωνώ απόλυτα ότι ήταν σημαντική αυτή η υπόθεση που αναφέρατε, όχι μόνο για την Ιταλία και την απόθεση, αλλά την απόθεση από τα σύνορα γενικά και την επιστροφή. Το έθεσα όταν επισκέφθηκα την Ιταλία και για τι ζωέ που χάνονται στη θάλασσα. Σχετική έκθεση διαπίστωσε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στην προστασία των ανθρωπίνων ζωών για ανθρώπου που ταξιδεύουν δια τη οδού και φτάνουν στι ακτέ τη Ευρώπη ή δεν φτάνουν στι ακτέ. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση, ένα ε, σημαντικό τομέα όπου εμεί και το Συμβούλιο τη Ευρώπη αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οδηγία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατήσουν παράνομου μετανάστε μέχρι 18 μήνε, να είναι σε κράτηση, είναι απάνθρωπο θεωρούμε, άσκοπο, αντιπαραγωγικό. Νομίζω ότι είναι ελάχιστο κοινό παρανομαστή, διότι η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέτρο τελευταίο έσχατο και μόνο εν ώψη απελάσεω. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, πόσοι παράνομοι μετανάστε απελάβνονται αφού έχουν κρατηθεί, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Άρα ε, υποφέρουν οι άνθρωποι άσκοπα ε, και είναι κάτι που απορρέει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει σε αρκετές ε, χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα, πολλά προβλήματα μάλλον. Όσον αφορά τη Ρωσία και την Τουρκία, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις, πολύ διαφορετικές. Αλλά υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ε, ομοιότητα. Έχουν υπουργού ε, δικαιοσύνη που είναι μεταρρυθμιστέ στο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται, αλλά εργάζονται υπό πολύ σοβαρού περιορισμού. Στη Ρωσία, παραδείγματο χάρη, όπω είπα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μα έδωσε πολύ καλή νομική βάση για διάλογο με τι ρωσικέ αρχέ και το Υπουργείο Δικαιοσύνη συγκεκριμένα και γνωρίζουν τα προβλήματα πάρα πολύ καλά και θέλουν να μειώσουν τον αριθμό υποθέσεων που πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να βρουν στο εσωτερικό ε, λύσεις. Τα προβλήματα στη Ρωσία, αλλά όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στην Ουκρανία και την Τουρκία επίσης, το πρόβλημα είναι, λέγω, όχι μόνο πολιτική παρέμβαση, αλλά και η στάση των εισαγγελέων, των δικαστών, που ενδιαφέρονται περισσότερο στην προάσπιση του κράτου ή αυτό που αντιλαμβάνουν σαν κρατικό συμφέρον, παρά να υπερασπιστούν τι ελευθερίε τι ατομικέ. Το είδαμε αυτό πρόσφατα στην περίπτωση Μαγνέτσκι, όπου αφού έκανε δήλωση ο κύριος Πούτιν, σταμάτησε ο εισαγγελέα τις κατηγορίες κατά κάποιου μέλους του ιατρικού προσωπικού που παρακολουθούσε την ιατρική περίθαλψη που χορηγείται στον κύριο Μαγνέσκι. Άρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσει και για εργασίες. Όσον αφορά την υπόθεση Μαγνίσκη, η εντολή μου δεν μου επιτρέπει να ασχολούμαι με άτομα, αλλά δείχνει πάρα πολύ καλά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει τονίσει την πτυχή της διαφθοράς και την ανάγκη που υπάρχει για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται αυτού του είδου τα ζητήματα. Εγώ εστιάζομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και εξετάζω τις συνθήκες κράτησης, ε, δικαιοσύνη που έχει χρειά πολιτική, ιατρική περίθαλψη, την ανάγκη να υπάρχει ε, κράτηση κατηγορουμένων πριν τη δίκη ε, και έχουμε την πολύ παράξενη υπόθεση των ποινικών κατηγοριών που απογγέλλονται κατά κάποιου ο οποίος είναι νεκρός. Πάρα πολύ παράξενη περίπτωση στην Τουρκία. προσβλέπουμε στην εφαρμογή του τέταρτου πακέτου δικαστικών μέτρων. Είμαστε στενή επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας. Ε, στην Τουρκία η κατάσταση περιπλέκεται από διάφορου παράγοντε, Από την ροή των Συρίων προσφύγων, με τη μάχη με το ΠΚΚ και τη σχέση που έχει με τι αρχέ που συνεχώ μεταβάλλουν τις σχέσεις, διάφορα πολιτικά ζητήματα. Ο προκάτοχό μου ετοίμασε μεγάλη έκθεση με θέμα το δικαστικό σύστημα διότι εντοπίσαμε ότι το δικαστικό σύστημα είναι το βασικό πρόβλημα όσον αφορά την ελευθερία του συναθρίζεστε, τη έκφραση. Οι δικαστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα φυλακίζονται και κρατούνται και ο Υπουργό Δικαιοσύνη είναι μεταρρυθμιστή όσον αφορά προσανατολισμό, αλλά πολύ συχνά συμβαίνουν πράγματα στο δικαστικό τομέα που είναι εκτό ελέγχου του. Έτσι θα έπρεπε να είναι πιθανότατα, αλλά μακάρι τα διαφορετικά τα πράγματα. Προτιθέμεθα να μεταβούμε εκεί και όχι μόνο να δούμε τι γίνεται στι προσπάθειε στο δικαστικό τομέα, αλλά να εξετάσουμε και τι νέε εξελίξει, τη δημιουργία του διαμεσολαβητή, του Εθνικού ε, Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι τουρκικέ αρχέ να προχωρήσουν σε αυτού του τομεί και να εξασφαλίσουμε ότι το τέταρτο αυτό πακέτο για το δικαστικό τομέα καλύπτει πολλέ από τι ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αντικατοπτρίζονται στι υποθέσει που είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Θεμελιών Δικαιωμάτων. Σαν την Τουρκία, ένα θέμα που δημιουργεί απογοήτευση, το άκουσα και από τον Υπουργό Δικαιοσύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν δημοσίευσε την έκθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση για το δικαστικό κλάδο όταν εξέταζε την κατάσταση στο δικαστικό τομέα και στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Αισθάνονται οι Τούρκοι λοιπόν ότι Υπάρχει μεγάλος φόρτος συναισθηματικός και πολιτικός αυτή τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωση Τουρκίας. Είπε όμως ότι θα τον βοηθούσε αν δημοσίευε η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διάφορες εκθέσεις για τον δικαστικό τομέα, την έκθεση screening, δίθηση ελέγχου των εξελίξεων. Όσον αφορά τους τσιγκάνους, τους Ρωμά και τις μειονότητες εν γέννη, στόχος μου δεν είναι να καλύψω ε, το έργο άλλων φορέων, αρμοδίων αλλά να προσπαθήσω να ενισχύσω τα διάφορα μηνύματα που στέλνουν οι άλλοι αρμόδιοι φορείς και στη σύμβαση πλαίσιο παροτρύνεται να επικυρώσουν αυτό το πλαίσιο οι χώρες όσες δεν το έχουν επικυρώσει για το ΕΚΒΙ θέλουμε γενικές στάσεις για την πολιτική να εξεταστούν από τις χώρες, να ληφθούν υπόψη και το ίδιο και με τη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τις ε, γλωσσικές μειονότητες το θέμα των Τσιγκάνων και των Ρωμά έχει αναδειθεί αρκετές φορές. Θα πρέπει να θεωρηθούν μειονότητα οι Ρωμά, αλλά ε, και σε άλλες χώρες και αυτό ισχύει και στην Τουρκία. Υπάρχουν θρησκευτικές μειονότητες εκεί που ε, θέλουν να έχουν αναγνώριση. Ε. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε και με την ύπατη ε, αρμοστία για τις ε, ουσικές μειονότητες πριν πάμε στη τεχική δημοκρατία και, στην, ε, και στο ΦΥΡΟΜ για να στέλνουμε παρεμφερή μηνύματα, τα ίδια μηνύματα όσον αφορά την παιδεία, την απομόνωση, το διαχωρισμό στην παιδεία, να βοηθήσουμε τους τσιγκάνους κλπ. Όσον αφορά τις άλλες μειονότητες, τις είδαμε στα πλαίσια τη καταπολέμησης τη διάκρισης. Σε ποιο βαθμό είναι αντικείμενο διάκρισης. πόσε πολιτικέ πολιτικές καταπολέμησης διάκρισης βοηθούν να πετύχουν πλήρη ισότητα στη χώρα που ζουν. Στη Ρωσία, πρόθεση όταν συνέστη όταν ετοιμάζω την έκθεση για τη δικαιοσύνη είναι να εξετάσω το τι γίνεται μετανάστευση. Προσελκύει η Ρωσία μετανάστες από τη γύρω περιοχή και είναι κάτι διαφορετικό από τι μειονότητε, αλλά υπάρχουν και κοινά σημεία. Στην Τουρκία ο μου ετοίμασε μεγάλη έκθεση όσον αφορά τι μειονότητε, εθνοτικέ και θρησκευτικέ, Πολλά από τα θέματα αφορούν την ελευθερία τη έκφραση και συνδέονται με του Κούρδους, με το κουρδικό ζήτημα. Όλα αυτά αναφύονται τακτικά. Η Ρώμα είναι η πιο πολύ συζητημένη υπόθεση αλλά και άλλε μειονότητε στα πλαίσια τη καταπολέμηση ε, των διακρίσεων. Δεν ξέρω αν απάντησα το ερώτημά σας, κύριε Κιγκεγκάλ, για τις μειονότητες και πώς αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των εργασιών μας. Uh, okay, και εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, είπατε δεν θέλετε να σχολιάσετε. Υποθέτω δεν έχετε κάποια προβλήματα σχετικά με αυτά που υπόθηκαν. Τα άλλο θέμα, περιπλοκότατο. Η πρόσβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πώ έχουμε προχωρήσει. Το θέτω σαν ερώτημα. Πώς έχουμε προχωρήσει εκεί. Πώς έχει προ... προχωρήσει η προετοιμασία. Δεν συσχετίζεται άμεσα με το έργο της Επιτροπής. Και έτσι λοιπόν μπορούσε να προβλεφθεί. Γνωρίζω ότι συνεχίζεται το έργο σας. Και είναι περίπλοκες και σύνθετες οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις. Και δεν θα μπορούσα να αυτό σχεδιάσω έτσι ε, των ενόντων. Τώρα, με ναι, και έχω τον λόγο, ε, δεν θα είχα κάτι το συγκεκριμένο να αναφέρω επ' αυτού. Δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένα θέματα που προετοιμάσαμε ως παρατηρήσεις. Σε ένα γενικότερο επίπεδο θα ήθελα να τονίσω αυτά τα οποία αναφέρθηκαν λέγοντας ότι εμείς συνεχίζουμε την συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και αυτό συμβαίνει και ακόμα και σε σχεδόν προσωπικό ή μη προσωπικό επίπεδο. Εμπλέκομαι και εμπλεκόμουνα στο έργο για την προπαρασκευή του στρατηγικού πλαισίου και το πρόγραμμα δράσης και τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου για τα δικαιώματα του ανθρώπου από πλευράς ΕΕ. Υπάρχουν αρκετές ανησυχίες που διατυπώθηκαν από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση τότε του Συμβουλίου της Ευρώπης για το αν θα υπήρχε κάποια ίσως επικάλυψη ή όχι αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις αρμοδιότητες και το έργο που αναπτύσσει ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο ειδικό εντεταλμένος της ΕΕ. Και η ίδια η εμπειρία, η πείρα μας κατέδειξε ότι δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχουν τέτοιες επικαλύψεις. Και αναφέρατε εσείς ε, και σε σχέση με τον Σταύρο Λαμπρινίδη τα θέματα ε, συνεργασίας σας. Νομίζω είναι ένα ευτυχές ε, παράδειγμα πώς μπορούν να συνεργάζονται με θετικό τρόπο τα δύο μας θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ cooperation να πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης γενικότερα. Νομίζω ότι ε, σε επιχειρησιακό επίπεδο, παραδείγματο χάρη πριν πάμε σε μια χώρα στα, δυτικά, Βαλκάνια ή στι χώρε τη Ανατολική ε, ε, εταιρική σχέση, είναι καλό ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και σε μερικέ χώρε είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε στα Δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολική εταιρική σχέση, γιατί οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, και σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, για την Τουρκία, για τη Ρωσία, ίσως είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Ε, γιατί εδώ υπάρχουν ε, κάποια θέματα που περιπλέκουν το δικό μου έργο ή το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για χώρες που είναι μέλη του. Με τον κύριο Λομπρινίδη είχα πολλές χρήσιμες ε, συναντήσεις και θα τον ξαναδώ σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι στις μεταξύ των χωρών εκεί όπου έχουμε κοινά θέματα στη μέση διάταξη η χώρα είναι η Ρωσία και έχουμε πολλά σημεία επί των οποίων συμφωνούμε για τη Ρωσία και θα περιμένω να δω πώς θα έχει ε, δημιουργήσει και εκείνο στο γραφείο του, γιατί εγώ είχα την πολυτέλεια να μπω σε μια υπηρεσία που λειτουργούσε ήδη, ενώ ο κ. Λεμπρινίδης έπρεπε να στήσει μια υπηρεσία εξ αρχή. Επομένω, περιμένω να δω το όραμα του κ. Λεμπρινίδη για το αντικείμενό του δύο θεματικά θέματα στα οποία επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό ε, ε, οι προτεραιότητέ μα είναι τα θέματα των ε, ομοφιλοφίλων, λεσβιών, διεμφυλικών κλπ. και τα θέματα διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτό αφορά όχι μόνο την Ρωσία αλλά και όλες τις χώρες του Συμβουλίου τη Ευρώπης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, και υπάρχει πεδίο συνεργασία και το διαδίκτυο θα αρχίσει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο έργο μας. Θα αρχίσουμε να παρακολουθούμε λεπτομερώς τις προσπάθειες των μεμονωμένων χωρών να, περιορίσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και θα εξετάσουμε επίσης ε, και θέματα απορρίτου και προστασίας δεδομένων και το πώς ορισμένες χώρες προσπαθούν ε, να ελέγξουν και να παρακολουθήσουν την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ε, κάποιες ερωτήσεις για τη ΦΥΡΟΜ και θα ήθελα να πούμε ε, κι εμείς ότι ετοιμάζουμε μια έκθεση. Ο κύριος Χάουιτ που είναι στη Σιέρα Λεόνε τώρα ετοιμάζει μια έκθεση για την ΦΥΡΟΜ και καλό θα ήταν να, ε, είμαστε σε επαφή. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη η έκθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και έχουμε και μια έκθεση για τη διαφθορά και τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα για χώρες εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης προγραμματίζουμε μια έκθεση για την ε, ελεύθερη άσκηση θρησκευτικών δικαιωμάτων και ελευθερία των πεπιθήσεων. Δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή. Εσείς είπατε ότι έχετε φοιτεία εξαετή. Εμείς έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές το 2014, οπότε μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει λίγο πολύ να έχουμε προχωρήσει. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε προχωρήσει σε όλα αυτά. Νομίζετε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή θα έχουν προστιθέμενη αξία αν συνεργαστούμε περισσότερο? Ξέρω ότι υπάρχει μια κοινοβουλευτική συνέλευση στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου συμμετέχουν βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επομένως μπορεί να μην είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι συμμετέχοντες. Να ξεκινήσω εγώ και μετά θα συμπληρώσει ο κύριος Πρέσβης. Όσον αφορά την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Περιμένουμε περίπου μία εβδομάδα μετά τις τοπικές εκλογές ε, για να εκδώσουμε την έκθεση και η έκθεση θα ασχοληθεί με δύο βασικά θέματα. Τους ε, Ρωμά και την, ε, το διαχωρισμό στην εκπαίδευση και το καθεστώς των απάτριδων και τις μετακινήσεις τους και επίσης ένα άλλο θέμα είναι η μεταβατική περίοδο για τη δικαιοσύνη εγκρίθηκε ε, κάποιος νόμος, πέρασε κάποιος νόμος ε, ιδιαίτερα ε, επίμαχος και η Επιτροπή της Βενετίας εξέθεσε, έκανε κάποια σχόλια με βάση και τη Συμφωνία της Αχρίδας. Τώρα, όσον αφορά την κοινοβουλευτική συνέλευση, όντως τα μέλη είναι βουλευτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται λιγότερο ή περισσότερο. Μερικοί είναι ιδιαίτερα δραστήριοι και κάνουν και πολλές εκθέσεις και έχουμε εισηγητές από πολλές χώρες και έχουμε και πολλές θεματικές ενότητες. Βέβαια, κάποιοι βουλευτέ ε, θεωρούν τη δική του χώρα ω προτεραιότητα, οπότε είναι λιγότερο δραστήριοι στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Έχουμε πολύ, πολύ καλού εισηγητέ για ορισμένα θέματα. Και θα δείτε ότι υπάρχει εισηγητή για τα θέματα των ομοφιλοφίλων ε, και ε, διεμφυλικών και για άλλα θέματα και όντως ε, αν έχετε κάποιο σχετικό θέμα μπορείτε να καλείτε τους εισηγητές κάθε φορά να σας κάνουν μια παρουσίαση για τη δουλειά που κάνουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να προσθέσετε εσείς κάτι? Ναι, κυρία Πρόεδρε. Uh, να σας πω ότι μια φορά το χρόνο γίνεται συνάντηση μεταξύ των Προεδριών των δύο εκλεγμένων φορέων της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στην τελευταία συνεδρίαση οι δύο πρόεδροι Ζαν Κλοντ Μινιού και ο Μάρτιν Σούλτ το Δεκέμβριο φέτος αποφάσισαν ότι θα αναθέσουν στο γενικό, στους γενικούς γραμματείς των δύο συνελεύσεων, των δύο φορέων, να ετοιμάσουν λεπτομέρειες για τακτικότερες επαφές και ανταλλαγή εκθέσεων και τεκμηρίωσης και για συνεδριάσεις, ως αυτό ενδείκνυται. Κυρίως εκθέσεις και επιστολές ετοιμάζονται στις δύο συνελεύσεις και αυτά τα έγγραφα είναι πολύ χρήσιμα για κάθε συνέλευση αντιστοίχως. Σας ευχαριστώ. Καλώς, λέει Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Δεν έχουμε τίποτα ε, που στο οποίο να διαφωνούμε βασικά όσον αφορά το περιεχόμενο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Καλό που σας ακούσαμε, ποιε είναι οι προτεραιότητές σας, ούτω ώστε να μπορούμε να ενισχύουμε ένα τον άλλον. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου των αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά μου έρχεται στο μυαλό ότι θεωρητικά οι περισσότερες αντιπροσωπείες της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν εστιακό σημείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όταν μιλάμε για Τουρκία και Ρωσία ε, είναι καλή πηγή πληροφοριών και είναι πολιτικά πιο εύκολο να οργανώνται συναντήσεις κλπ. Θα τα ξαναπούμε στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες ίσως θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι τακτικά στις Βρυξέλλες. Με τα χαράς. Να συναντηθούμε, έρχεστε και εσείς τακτικά στο Στρασβούργο. Με τα χαράς λοιπόν να συναντηθώ μαζί σας όποτε σας βολεύει. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τουρκία συναντήθηκα με το κεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης. Στο ΦΥΡΑΜ, ΦΥΡΟΜ συναντήθηκα με όλου του της τη Ευρωπαϊκή Ενώση, την αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Έχουμε καλές επαφές με την Υπηρεσία εξωτερικής δράσης και νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η επαφή, διότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να μάθουμε ένα από τον άλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστήκη πρόεδρος. So uh, let us continue um, Συνεχίσουμε τώρα. Ελπίζω ότι λειτουργούν τεχνικά όλα τα μέσα. Λοιπόν, τώρα παρακαλώ ησυχία και καθίστε αν θέλετε. Τώρα έχουμε και την ακρόαση για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία. Συζητώντας αυτό το θέμα στο διευρυμένο Προεδρείο όταν το συζητήσαμε, είδαμε ότι είναι ακαθόδες περίπλοκο θέμα, όχι μόνο λόγω του ότι είναι δυσχερέστατη η κατάσταση στην ίδια τη Συρία, αλλά και επειδή διεθνώς οι κατευθυντήριες γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο θεσπίστηκαν και εγκρίθηκαν μεν, όμως ουσιαστικά εμείς δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι γίνεται και διαπιστώσαμε εμείς αυτό στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή οι παρόντες και Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι ΜΚΟ, ιδιαίτερα η Amnesty International, ζήτησαν από την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου να καθοδηγήσει το, ε, την ομάδα ε, του Συμβουλίου ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που ε, παρουσιάζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ετήσιο φόρουμ το 2011. Ξεκινήσαμε με συζητήσεις λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη Συρία και μάθαμε ότι υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος της συζήτησης για το πώς εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις, ε, αυτούς τους προσανατολισμούς της ΕΕ. Στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να διεξαγάγουμε αυτή την ακρόαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης, την κυρία Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, κυρία Εύα Ζολή. Σας ευχαριστούμε καλώ ήρθατε και θα, έχετε, έτσι, θα υπάρχει ευδιάκριτο ρόλο για το τι μπορούμε να πράξουμε εμεί. Έχουμε κάποιες συναντήσεις ε, από κοινού, αλλά γενικά Επιτρέψτε μου να πω ότι στην ε, Επιτροπή, μα μας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντιμετωπίζουμε συνολικά όλες τις περιπτώσεις ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και έχουμε ε, ιδιαίτερη επικέντρωση στο μείγμα μεταξύ των πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και νομίζω είναι μια σωστή ε, ισορροπημένη προσέγγιση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εχθές είχαμε και την κατάσταση της Ρωσίας που συχνά εγγράφεται στην ημερήσια διάταξή μας και εστιαστήκαμε ιδιαίτερα για το πώς η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τους φτωχούς, ε, τους ε, ανεχείς πολίτες στην Ρωσία Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, αλλά έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και πολιτικών, παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων επίσης. Είναι πληρέστατη η ημερήσια διάταξή μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα θέλατε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με τα χαρά ε, συμπροεδρεύω σε αυτή τη δημόσια κρόση σήμερα την κοινή κρόση των δύο επιτροπών μας, ακόμα και αν τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι πολύ δραματικά και οι περιστάσεις όσον αφορά το θέμα αυτό, η κατάσταση στη Συρία, ε, είναι φρικτή η κατάσταση στη Συρία. Εδώ και δύο χρόνια δεν μπορούμε παρά διαπιστώνουμε την αδυναμία μας της τραγωδίας της που λαμβάνει η χώρα στη Συρία που έχει οδηγήσει σε πάνω από 60.000 νεκρούς σύμφωνα με την υπατιαρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πολιτική κατάσταση γίνεται, ε, η λύση πολιτική μάλλον γίνεται όλο και πιο δύσκολη κάθε μέρα. Πρέπει να αρκεστούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, στο να δείξουμε την αλληλεγγύη προς το Συριακό λαό μέσω ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμα και γενναιόδορη αν είναι και αποτελεσματικότατη αν είναι, δεν μπορεί να επιλύσει από μόνη την ανθρωπιστική κρίση που σημειώνεται επιτόπου και στη Συρία και πέρα από τα σύνορά της όμως και επιδεινώνεται καθημερινά χωρίς να φαίνεται να είναι κοντά καμία λύση όπως μας το είπε με θλίψη και πίκρα η Ευρωπαϊκή Επίτροπος ε, που είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια η κυρία Κρυσταλίνα Ζιόρζεβα στην Επιτροπή Ανάπτυξης την περασμένη Δευτέρα. Έτσι δε περαιτέρω όταν οι θεμελιώδεις αρχές ε, δέχονται επίθεση 15 ανθρω... εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια έχασαν τη ζωή τους στη Συρία και ανθρωπιστικές εφοδιοπομπές ε, δέχονται επιθέσεις και πυροβολισμούς τακτικά. Ξέρουμε ότι τα νοσοκομεία ήταν στόχοι ε, βομβαρδισμών. Η πρόσβαση του Συριακού στους στο πληγέντα πληθυσμό της Συρίας γίνεται όλο και πιο δύσκολη, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας Μία αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια δεν καθορίζεται μόνο από την επαρκή χρηματοδότηση. Πρέπει να σας πω ποια είναι η ανησυχία μου όσον αφορά ότι είναι στα μισά πλέον το απόθεμα. Μειώθηκε στα μισά η χρηματοδότησή μας σύμφωνα στις τελευταίες συμφωνίες για την πολιτική χρηματοδότηση. Το μισό κονδύλι έχουμε. Λοιπόν, χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική είναι η απεριόριστη πρόσβαση στον ευάλωτο πληθυσμό και να ε, γίνονται σεβαστοί από όλα τα μέρη οι κανόνες για την ε, συνθήκες χορήγηση ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ των θεμελιωδών αρχών των ανθρωπιστικών, ανθρώπινη προσέγγιση, αμεροληψία, ανεξαρτησία στην προσέγγιση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτές οι αρχές εντάσσονται στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και είναι στεμελιώδεις αρχές για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορείς για την ανθρωπιστική βοήθεια που παίρνουν τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα να μπορούν να λειτουργούν επί τόπου μέσα σε πλαίσια ασφαλείας και θέματα πολιτικά ε, περίπλοκες συνθήκες όπως είναι στην ε, Συρία. Χρειάζεται συνένεση ευρωπαϊκή για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, υπάρχουν και έγγραφα αναφορά που έχει υπογράψει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη για ανθρωπιστική βοήθεια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν υπογραφεί ε, έγραφα το 2007. Η αρμόδιο επίτροπο μα διαβεβαίωσε ότι ε, η ανθρωπιστική βοήθεια δίδεται σύμφωνα στι ανθρωπιστικέ αρχέ. Πολιτική απόλυτη ουδετερότητα ακολουθείται προ όλα τα μέρη. όσον αφορά την κατάσταση Συρία, η επίτροπο ε, είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε να μην δώσουν πολιτική χρειά στην ανθρωπιστική βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διότι αυτό θα ήταν ει βάρο των φορέων που προσπαθούν επιτόπου να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια. χρειάζεται η βοήθεια να φτάνει σε αυτού που την έχουν ανάγκη ανεξάρτητα που ε, βρίσκονται σε περιοχέ που ελέγχονται είτε από του επαναστάτε είτε από την κυβέρνηση. Ο Ζαν Λουίντε Προβέρ, ο εισηγητή μα, μάλλον που είναι διευθυντή γενική Διευθύνσεω ΕΚΟ, μπορεί να μα πει περισσότερε λεπτομέρειε για τις συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά το να γίνονται σεβαστά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κατάσταση αυτή που είναι περίπλοκη στη Συρία. Ο κύριος Ντεπχαβέρ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι διευκολύνεται σημαντικά το έργο μου σήμερα το πρωί σε σχέση με την παρουσίαση που έγινε από το, την επικεφαλής ε, μου την Επίτροπο κυρία Γεωργίεβα και που με ιδιαίτερα εύγλωτο τρόπο υπενθύμισε ποια είναι τα κύρια μηνύματα και τα κύρια μελήματα από πλευράς μας προσπαθώντας σε μια καθημερινή βάση να ανταποκριθούμε με, έναντι αυτών που είναι σίγουρα η χειρότερη και μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που βιώσαμε και βιώνουμε. Είναι σαφέστατο παράδειγμα σήμερα η Συρία. Τι μπορεί να συμβεί όταν τα δικαιώματα του ανθρώπου συστηματικά παραβιάζονται ξεκινώντας με διαδηλώσεις πριν από δύο χρόνια. Σήμερα αυτά είναι μια έκδηλη κρίση εκατομμυρίων ανθρώπων που χρειάζονται άμεση βοήθεια, δύο εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων λιγότεροι από 900.000 οι πρόσφυγες συνολικά και το αναφέρατε και εσείς και είπατε ότι όλες οι προβλέψεις για το αν είναι δυνατόν να υπάρξουν και όλα τέτοιου είδους προβλέψεις σε σχέση με μια τέτοια χαοτική κατάσταση μας οδηγούν στο να σκεφτόμαστε σήμερα υπό τους όρους ε, της Δευτέρας Παρουσίας, μιας πραγματικής συντέλειας του κόσμου σε σχέση με την κατάσταση που είναι δραματική εκεί, χωρίς καμιά ελπίδα. Είναι μακρότατος ο κατάλογος ε, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ε, τέτοιου είδους ομοτήτων και σε σχέση και με την, ε, τις διακριβώσεις που οι τελευταίες είναι μέχρι και την 18η Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά τι δείχνει δείχνουν όλα αυτά. Αυτή η έκθεση τονίζει με κάθε τρόπο το γεγονός ότι έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, φρικαλαιότητες και παραβιάσεις ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και από τις δύο πλευρές, και από τους αντάρτες και από τις κυβερνητικές δυνάμεις εγκλήματα τα οποία έχουν ε, σημειωθεί παρότι και από τους αντάρτες σε μικρότερο βαθμό από ό,τι σε σχέση με τα, ε, τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις. Η Διεθνής Επιτροπή, Εξεταστική Διεθνής Επιτροπή συνιστά ότι θα πρέπει το Συμβούλιο το Ασφαλείας των ΗΠΑ Εθνών να αναλάβει άμεσα δράση όσον αφορά την προσαγωγή ή δυνατόν των υπευθύνων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εδώ έγκυται ακριβώς το πρόβλημα. Το να βλέπει κανείς ότι δεν ήταν σε θέση το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών να ομιλήσει με μια κοινή φωνή επ' αυτών των θεμάτων, όχι μόνο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά σε εισαγωγικά και σε όσον αφορά απλά σε εισαγωγικά θέματα. Θεμελιώδους σημασία θέματα όσον αφορά την πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ λοιπόν και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο και ε, επανειλημμένα έχει ε, διατυπώσει έκκληση για το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του, ανθρωπιστικού διεθνούς ε, δικαίου ακόμα και την Δευτέρα αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο αυτή η έκκληση. Και με το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών που έχει τροχοπεδηθεί πιστεύουν πολλοί ότι δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή που έχει καταλήξει σε μια ανθρωπιστική κόλαση και μια ε, κατάσταση στη Συρία. Και σε σχέση με το ανθρωπιστικό αυτό πλαίσιο ανθρωπιστικού δικαίου τα προσκόμματα που υπάρχουν και ιδίως η έντονη βία έχουν καταστήσει ανέφικτο στους εμπλεκόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους και ιδιαίτερα με τον επιταχυνόμενο αριθμό όλων και περισσότερων θυμάτων από πλευράς στατιστικής. Ε, βλέπουμε ότι γεωμετρικά αυξάνονται οι ανάγκες, ενώ η βοήθεια που μπορούμε να παράσχουμε μόνο με πολύ μικρό και βραδύ ρυθμό μπορεί να αυξηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί όλους τους να παράσχει αυτή την σύνδρομή μας, να δώσουμε τη βοήθειά μας με κάθε τρόπο, με ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ωστόσο αυτό δεν είναι ούτε και απλό, ούτε και απόλυτα αποτελεσματικό σε αυτή τη φάση δεδομένων αυτών των περιορισμών και ε, ούτως εχόντων των πραγμάτων. Θα έπρεπε να υπάρχει ή η συνένεση και των κυβερνητικών δυνάμεων ή και των αντατών ή αμφωτέρων. Ωστόσο, οι αντάρτες δεν έχουν μια ενιαία ε, εναρμονισμένη δομή. Ή θα πρέπει επίσης να χρειάζεται και η συνένεση επιπλέον ομόρων γειτονικών κρατών Όλα, όλες αυτές οι χώρες είπαν τουλάχιστον επίσημα ότι δεν προτίθενται να παραβιάσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ε, Συρίας και να αναμειχθούν. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί, όπως γνωρίζετε, στην κατάσταση όπως επικρατεί σήμερα στη Βόρεια Συρία. Η κατάσταση είναι πολύ αρνητική. Ωστόσο, δεν είναι τόσο κακή ή αρνητική ή χειρότερη, σε χειρότερη ακόμα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Στο βορρά της Συρίας ε, βλέπουμε έντονες, ε, έντονη ανάγκη να ε, συνδράμουμε και να βοηθήσουμε να σωθούν ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε αντίσκηνα κατά μήκος των τουρκικών συνόρων πολλοί άνθρωποι που έχουν καταφύγει εκεί και έχουμε άμεσο πρόβλημα προσπελασιμότητας, πρόσβασης ε, αυτών των ε, ανθρώπων στις ε, να καλυφθούν οι κυριότερες ανάγκες τους. Ένα από τα κεκτημένα δεν πρέπει να το υποβαθμίσουμε είναι η ανάπτυξη εγκάρσεων ε, δυνατοτήτων επαφών με αυτοκινητοπομπές ε, από πλευράς μας ώστε να καταλήξουν τα υλικά και η βοήθειά μας στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στο βορρά της Συρίας. Είναι συμβολικά και αξίζουν να αναφερθούν όλα αυτά. Όμως όλα αυτά είναι περιορισμένης εμβέλειας και δεν είναι αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται για να καλύψουμε τις ανάγκες σε ευρύτερη κλίμακα μιας τέτοιας ανθρωπιστικής έκδηλης κρίσης. Και για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους πρέπει να πω και να τονίσω ότι οι διεργασίες, οι ε, διαδικασίες, ε, οι, τα όσα γίνονται για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους πραγματικά μας κάνουν να βρισκόμαστε σε απόγνωση, να απογοητευόμαστε λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν ε, να, βοηθήσουν τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε. Το να παράσχουμε αυτή την σημαντικότατη βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται άμεσα αυτή τη βοήθεια μπορείτε όλοι να φανταστείτε ότι είναι η ανώτατη πρώτη προτεραιότητά μας. Θέματα προστασίας έχουν την κυριότερη σημασία. Με όλες τις εκθέσεις που αναφέρουν γεγονότα βίας εις βάρος γυναικών, την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού έχω υπόψη μου για την βία εις βάρος των γυναικών και φυσικά και τις εκθέσεις όσον αφορά διάκριτέ δολοφονίε και φρικαλαιότητες. Και εδώ πάλι αναφέρομαι στη Διεθνή Επιτροπή ε, Διακρύβωσης στην έκθεση που συνέταξε ολοκληρώνοντας αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις ε, θα έπρεπε να επαναλάβω και να τονίσω ότι όλα αυτά τονίζουν για άλλη μια φορά ότι έχουμε πραγματικά μια de facto ατιμορρησία όσων διαπράττουν εγκλήματα και παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτή η ατιμορρησία θα οδηγήσει στην αύξηση και επιδείνωση των ε, γεγονότων αυτών ε, και της κατάστασης αυτής. Τη απουσία οποιασδήποτε δράσης από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών λοιπόν επανειλημμένα και διαρκώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους συμβάντα και μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανθρωπιστική συνδρομή, το διεθνές ανθρωπιστικό πλαίσιο ως ανθρωπιστικό δίκαιο, θα μπορούσαν όλα αυτά να αποτελούν ένα, ένα στοιχείο που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τα δεινά που υφίσταται ο λαός της Συρίας και θα μπορούσαν να, αν είχαμε και την ε, περαιτέρω σύνδρομη των ε, ε, αποτελεσματική σύνδρομη να καλύψουμε τις κατεπίγουσες ανάγκες που θα αυξάνονται διαρκώς και όπως γνωρίζουμε θα αυξηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες αλλά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε το λόγο στον πρέσβη από την Ελβετία να ευχαριστήσω την Ελβετία για αυτή την πρωτοβουλία σε διαφορετικά επίπεδα. Προσπαθείτε να βοηθήσετε την κατάσταση στη Συρία. Λοιπόν, θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την επόμενη εβδομάδα και βασική μέρη της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η Συρία. Και αυτό το ψήφισμα έμαθα ότι ατυχώς δεν έχει κοινή θέση. Όλα τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν να υποστηρίξουν αυτό το, αυτή την πρόταση. Μόνο μία χώρα διαφωνεί. Καλή η πρωτοβουλία, δουλεύετε ε, και προσπαθείτε να, να αλλάξετε γνώμη και να μας στηρίξει και τελευταία χώρα η Σουηδία. Δεν ακολουθεί τη λογική της συνήθους πολιτικής ε, της ε, Σουηδίας που συνήθως ακολουθεί διαφορετική πορεία μέχρι τώρα. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Πρέσβη. Θα μιλήσετε και για το ελβετικό, για την Ελβετική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά και η Διεθνή Επιτροπή και πώς θα μπορούμε να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση γενικά στον κόσμο με, τα, με τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για αυτά που είπατε για το τι έχει κάνει η Ελβετία στο πλαίσιο της παραπομπής της κατάστασης της Συρίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κυρία, Επίτρο... Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης, ε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά το ότι μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή την μεικτή ακρόαση για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Με μια μεικτή ακρόαση δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών και εκ μέρου τη ελβετική κυβέρνηση θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω για την κοινή πρωτοβουλία της Ελβετίας και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την συμβατότητα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, κάτι που ξεκινήσαμε πέρυσι ως συνέχεια της 21ης συνάντησης ε, του ε, Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Σιμισελίνου. Ε, έχουμε μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Συρία και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελβετία ελβετική πρωτοβουλία του, ε, της Επιτροπής ε, του Ερυθρού Σταυρού δεν θα πρέπει να συσχετιστεί με συγκεκριμένες σειράξεις, ούτε με την κατάσταση στη Συρία, ούτε με καμία άλλη χώρα. Παρόλα αυτά είναι προφανές ότι οι πολλαπλές ε, ένοπλες σειράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο μας απασχολούν ε, και βρίσκονται πίσω από τέτοιες προσπάθειες. Ε, η Ελβετία είναι υπέρ ε, της, του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε τέτοιες σειράξεις και είμαστε κατά της ατιμορρησίας για εγκλήματα πολέμου. Αρκεί λοιπόν να αναφέρουμε ότι κατόπιν πρωτοβουλία της χώρας μου, μία επιστολή που συνυπεγράφει από περίπου 60 χώρες, εστάλει ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 14 Ιανουαρίου και ζητάμε να αναφέρονται ε, τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν στη Συρία ε, και να σταλούν ε, ε, στην εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του χάρτη. Ε, η Συρία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Συμβουλίου Υπουργών των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας σε σχέση με αυτή την επιστολή που στείλαμε πρωτοβουλία της Ελβετίας ε, στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Κυρίε και κύριοι, την περασμένη Κυριακή στις 7 Φεβρουαρίου η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού που ιδρύθηκε το 1863 από πέντε Ελβετούς πολίτες από τη Γενέβη εόρτασε την 150η της επέτειο, πριν από πέντε μέρες δηλαδή. Και ε, η διεθνής κοινότητα του χρόνου θα εορτάσει την έγκριση της Σύμβασης της Γενέβης του 1864, που είναι η πρώτη σύγχρονη συνθήκη για το ανθρωπιστικό δίκαιο. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο είναι ένα σημαντικό επίτευγμα του πολιτισμού μας. Οι ένοπλες σειράξει είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με την ανθρώπινη ύπαρξη και θα πρέπει να φροντίζουμε ε, να αποφεύγονται ε, ταλαιπωρίες που μπορούν να αποφεύγονται και να μην ε, εκπίπτουμε σε βαρβαρότητες. Θα πρέπει μέσω αυτού του νομοθετικού μέσου να δίδονται τα μέσα για να αποφεύγονται οι παραβιάσεις του δικαίου και δεύτερον σε περιπτώσεις που υπάρχουν παραβιάσεις να λαμβάνονται μέτρα για να σταματούν αυτές οι παραβιάσεις. Και τρίτον, θα πρέπει να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι κάθε φορά για τις παραβιάσεις. Και όσον αφορά την πρόληψη και όσον αφορά την καταστολή, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο ε, τα τελευταία χρόνια Όσον αφορά όμως ε, την πάυση των παραβιάσεων, η κατάσταση ε, δεν είναι ικανοποιητική ακόμη. Ακόμη και 150 χρόνια μετά την κωδικοποίηση του διεθνούς, ε, από τότε που ξεκίνησε η κωδικοποίηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν το έχουμε επιτύχει. Πάντοτε οι ένοπλες σειράξεις είναι βασική πρόκληση για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Είναι ανησυχητική όμω ε, η αδιαφορία προ τι αρχέ του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Παραβιάζεται καθημερινά και από κρατικέ ένοπλε δυνάμει και από μη κρατικέ ένοπλε ομάδε. Και οι παραβιάσεις ε, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ε, δημιουργούν προβλήματα και στους μαχόμενους αλλά και στον άμαχο πληθυσμό. Μας ανησυχεί λοιπόν και η κατάσταση στη Συρία για αυτούς τους λόγους και διότι ε, αυτό σημαίνει ε, σημαντικά προβλήματα για τους ε, πολίτες και τους εμπλεκόμενους, αλλά και διότι πλήττεται το κύρος του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Τα περισσότερα ανθρωπιστικά προβλήματα δεν θα υπήρχαν αν ε, γινόταν πλήρως σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο από τα διάφορα μέρη. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας, αλλά η αδιαφορία. Οι κανόνες υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι δεν τηρούνται. Χρειάζεται λοιπόν να θεσπίσουμε όχι νέους κανόνες, αλλά μέτρα για να τηρούνται καλύτερα και να εφαρμόζονται καλύτερα οι σχετικές διατάξεις. Οι συμβαλόμενοι στη Σύμβαση της Γενέβης και στο Πρωτόκολλο 1 έχουν συμφωνήσει με κάποιους ε, μηχανισμούς. Είναι ένας μικρός αριθμός μηχανισμών που θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Δεν ε, ανταποκρίνονται όμως στη σημερινή πραγματικότητα, διότι δεν σχεδιάστηκαν για ένοπλες σειράξεις που δεν είναι διεθνείς. Αυτές ε, οι ένοπλες σειράξεις είναι, αποτελούν την ε, πλειοψηφία σήμερα. Άρα τα μέσα που έχουμε στη, ε, διάθεσή μας δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι σε περίπτωση ένοπλης σύραξης δεν μπορούμε να έχουμε την συνένεση όλων των εμπλεκομένων θα έπρεπε όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμπεριλαμβάνονται σε ένα σύστημα στο οποίο και θα ανταποκρίνονται. Γι' αυτό δεν είναι λειτουργικό το σύστημα αυτό και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται πλέον. Και υπάρχει και άλλη μία δυσκολία όσον αφορά την τήρηση της Σύμβασης της Γενέβης. Το Παγκόσμιο Φόρουμ στο οποίο μπορούν να συναντηθούν και να συζητηθούν, να συναντηθούν οι εμπλεκόμενοι και να συναντηθούν, είναι η διεθνή διάσκεψη του διεθνού Ερυθρού Σταυρού και τη Ερυθρά ε, Ημισελίνου. Έχει τεράστια σημασία για τα ανθρωπιστικά θέματα γενικότερα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια διάσκεψη γίνεται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια. Και υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα έπρεπε τα διάφορα κράτη να μπορούν να συζητούν πολύ πιο συχνά και όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και όσον αφορά την συμμόρφωση. Είναι ιδιαίτερα προβληματική η τωρινή κατάσταση και ενδέχεται να κλιμακωθεί αρνητικά και να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αδιαφορία από τις διάφορες χώρες, πράγμα το οποίο θα διαβρώσει την αξιοπιστία αυτού του θεμελιώδους ε, δικαίου. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Δεν υπάρχει μια εύκολη λύση στην τωρινή νομική κατάσταση. Οι χώρες δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ακόμη και αν θα το επιθυμούσαν διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Υπάρχει ένα κενό λοιπόν στη συμμόρφωση, πράγμα που μας έχει οδηγήσει στην κατάσταση όπου οι θεσμοί που δημιουργούνται ε, στο πλαίσιο διαφορετικών μορφών δικαίου εστιάζονται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια θετική ανάπτυξη, αλλά δυνητικά και αυτό είναι προβληματικό όσον αφορά την αποδοχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τους βασικούς εμπλεκομένους η 31η διάσκεψη Ερυθρού Σταυρού Θέση Μισελίνου το Δεκέμβριο του 2011 τόνισε τη σημασία του να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συμμόρφωσης και να εντοπιστούν τρόποι για να ενισχυθεί ο διάλογο ε, μεταξύ των κρατών για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ακόμη αναφέρεται ότι θα πρέπει οι συστάσεις να υποβληθούν στην 32η διάσκεψη που θα γίνει το 2015. Στη συνέχεια αυτών, η Ελβετία και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησαν μια διαδικασία για να προσφέρουν ε, στι διάφορες χώρες ευκαιρίε ε, να ε, ενισχύσουν τη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο είναι παγκόσμιο και οι χώρες είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνε να διασφαλίσουν την τήρηση του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Επομένω, το θέμα τη ενίσχυση τη συμμόρφωσης αφορά όλε τι χώρε. Και επομένως η διαδικασία την οποία ξεκινήσαμε θα πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής και πολυσυλλεκτική, ούτως ώστε όλες οι χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της συμμετοχής όλων, οργανώσαμε την πρώτη συνάντηση χωρών στη Γενέβη πέρυσι τον Ιούλιο. Και θέλουμε να συνεχίσουμε και να οργανώνουμε ετησίως τέτοιες συναντήσεις από τώρα μέχρι το 2015. Όταν αναλύουμε τους λόγους για την ευρύτερα διαδεδομένη μη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, βλέπουμε ότι τα εξή θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτον, οι χώρες που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνε για την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη συζήτηση για την ενίσχυση της συμμόρφωσης και χρειάζεται για αυτό το λόγο ένα κατάλληλο διεθνές φόρουμ. Δεύτερον, ε, επειδή οι φυστάμενοι μηχανισμοί συμμόρφωσης με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν πληρούν το στόχο τους, θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να τους ενισχύσουμε ή για να τους συμπληρώσουμε ή ενδεχομένως θα πρέπει να σκεφτούμε τη δημιουργία κάποιου νέου μέσου. Τρίτον, Μία ειλικρινής ανάλυση των λόγων για τη δυσλειτουργία του τωρινού μηχανισμού συμμόρφωσης καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει ένα συνεκτικό σύστημα που να έχει συνιστώσεις που αλληλοσυνδέονται, ούτως ώστε να ανταποκρινόμαστε με την απαραίτητη ευελιξία στις ε, δεδομένες προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι μετά από 150 χρόνια το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ακόμη δεν έχει αποτελεσματικά εργαλεία για να διασφαλίσει ότι τα κράτη θα συμμορφούνται με τις υποχρεώσεις τους σε καιρό ειρήνης, πόσο μάλλον σε καιρό πολέμου, μας δίνει μια πρόγευση του δύσκολου έργου που μας περιμένει. Δεν υπάρχει λοιπόν μια εύκολη λύση για τα προβλήματα που σας προανέφερα. Αντιθέτως, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μιας πολύπλοκης διαδικασίας που θα απαιτήσει χρόνο, ενδεχομένως αρκετά χρόνια, μέχρι ότου υπάρξουν αποτελέσματα. Και για να υπάρξουν αποτελέσματα θα πρέπει τα κράτη να αναπτύξουν, να ευαισθητοποιηθούν για τις διαστάσεις του προβλήματος της μη συμμόρφωσης. Και αυτή η ευαισθητοποίηση είναι ο πρώτος ενδιάμεσος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ένα απαραίτητο προαπαιτούμενο για να αναπτυχθεί η κατάλληλη δυναμική που θα φέρει και τις λύσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Ambassador Lang. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη Λάγκ. Κύριε Λάγκ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Λέτε ότι υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δίνουμε το λόγο, βλέπετε τώρα, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βλέποντας πόσο συχνά συζητάμε τι κατευθυντήριε γραμμέ Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το κάνουμε συχνά. Είναι η πρώτη φορά που από κοινού κοιτάμε αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ για το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο κ. Φάνα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα ήθελα να μας πει πώς αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές υλοποιούνται. Διότι εκεί λέγει, σε αυτές τις γραμμές που θετήθηκαν εν έτη 2009, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρεώσει τώρα να προωθεί τη συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο με ορατό και συνεπές τρόπο και να διαθέσει ε, τα κατάλληλα ε, επιχειρησιακά εργαλεία. Σαν κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσουμε να μας πει εξωτερική υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πώς αυτή η δέσμευση υλοποιείται στο έργο σας. Κύριε Σουόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ο κύριος με ιδιαίτερα ευγωτό τρόπο μίλησε για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ανθρωπιστική καταστροφή έκδηλη σήμερα στη Συρία ενώπιόν μας. Τα μελήματα και ανησυχία της ΕΕ σε σχέση με τη Συρία έχουν νομίζω επαρκώς και με καλό τρόπο καταγραφεί. Δίνοντας συνέχεια λοιπόν στην ερώτησή σας κυρία Πρόεδρε για το πώς η τη γραμμές ΕΕ όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ω πλαίσιο φυσικά διαφορετικό από το ανθρωπιστικό δίκαιο αφιευτού εφαρμόζονται και υλοποιούνται θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας και δίνοντας συνέχεια στην παρατήρηση του πρέσβεως Λάγκ για την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για να διασφαλίσουμε την ε, συμμόρφωση σε σχέση με αυτά. Και ως πρώτη παρατήρηση από πλευράς μου θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι σαφές υπό το πρίσμα της ΕΕ ότι το, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο υπερβολικά συχνά αποτελεί αντικείμενο παραβιάσεων και γι' αυτό παρακολουθεί εκ του σύνεγγης, ιδιαίτερα εκ του σύνεγγης ΕΕ τα τεκτενόμενα και αποκοινούμε την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προσβλέπουν στη δημιουργία ενός μηχανισμού ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο αυτή είναι η κυριότερη σημερινή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και η ΕΕ είναι υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλίας και προσπάθειας ώστε να διασφαλιστεί λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις και να τερματιστεί επιτέλους η ατιμορρησία όσον αφορά την, τέτοιου είδους εγκλήματα και παραβιάσεις. Και να εξεταστεί το εφικτό της ε, θεσμοθέτησης της δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ως προς την ε, επίτευξη αυτών των στόχων. Άμεσα όμως το άμεσο μέλλον, επειδή αυτό μπορεί να είναι ένας απότερος στόχος και να χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα, πράττει ε, σχεδόν αρκετά πράγματα η ΕΕ και μέσω τριών κυρίων αξώνων, ζητώ συγγνώμη για την βραχνάδα μου, Um, Και... θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας, τονίζοντας από πλευράς μου το ότι στον τομέα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας είναι περιορισμένες. Είναι τα κράτη-μέλη τα ίδια και όχι τόσο ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προσυπογράψει τις τέσσερις ε, συμβάσεις και συνθήκες της Γενέβης και τα πρόσθετα πρωτόκολλα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι εκείνα τα οποία δίνουν συνέχεια σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και υλοποιούν τέτοιες δράσεις. Φυσικά υπάρχει και ένας ρόλος από πλευράς μας για να συντονίζεται ε, ως ε, καταλήτης, ας το πω έτσι, η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου στην πρακτική εφαρμογή όλων αυτών. Εξού και αντανακλώνται αυτά τα στοιχεία στο στρατηγικό πλαίσιο, στο πρόγραμμα δράσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου που εγκρίναμε πέρυσι. Έτσι λοιπόν η αρχηγοί επικεφαλής ε, αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπρόσωποι, οι ειδικοί εντεταλμένοι όλοι με αυτές τις απαιτήσεις πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις για οποιασδήποτε παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου διαπιστώνουν και να υποβάλουν συστάσεις για την ανάληψη ε, αντίστοιχα αποτελεσματικής δράσης. Έχουμε λοιπόν αυτά τα μέσα στη διάθεσή μας και τον ε, διάλογο, τα διαβήματα, ε, δημόσιες δηλώσεις ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους παραβιάσεις αποτελεσματικά και επιπρόσθετα η προσανατολισμοί, οι κατευθυντήριες γραμμές που πρώτα ε, υιοθετήθηκαν το 2005 και αναθεωρήθηκαν το 2009 υπογραμμίζουν την σπουδαιότητα του θέματος της λογοδοσίας που πρέπει να διασφαλίζεται για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και υπογραμμίζει αυτό την συνεκτικότητα ε, και συνέπεια από πλευράς μας όσον αφορά το διεθνές ε, ε, δικαστήριο που πρέπει να επιλαμβάνεται τέτοιων περιπτώσεων. Και αναφερόμενο στις δραστηριότητές μας, η πρώτη αντανακλάτε στις δεσμεύσεις ε, και στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τα κράτη-μέλη κατά την 31η Διεθνή Σύνοδο των, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Ένα τέτοιο ήταν αίτημα όλα τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν όλα τα μέσα που αποτελούν στοιχεία πυρήνα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού που ακόμα δεν έχουν ε, προσυπογράψει ή δεν έχουν επικυρώσει ώστε μέχρι την επόμενη ε, διάσκεψη το 2015 να έχει ολοκληρωθεί και ε, το έργο για την ε, επιτέλεση αυτού του στόχου βρίσκεται υπό εξέλιξη και προοδεύουμε η Φινλανδία ή η Πολωνία επικύρωσαν την σύμβαση της Οτάβας για την ε, ε, μεταφορά και ε, χρήση των και εξουδετέρωση των ναρκών προσωπικού. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν προσυπογράψει αυτή τη σύμβαση και έτσι λοιπόν μπορεί με μεγαλύτερο κύρος και αποτελεσματικότητα να ακολουθήσει την επίτευξη αυτών των στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά διαβήματα εναντί τρίτων χωρών έχουν έχουν ε, ε, λάβει χώρα και έχουμε και εξτρατήσει υπεραιτέρω διαβήματα όσον αφορά την τύχη αυτή. Κάθε έτος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλει σημαντικές δηλώσεις προς αυτά. Η πιο πρόσφατη της 17ης Φεβρουαρίου για την 150η επέτειο της ε, ίδρυσης ε, του ε, εγκαθίδησης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Δεύτερον, μια νέα προώθηση, όθηση δόθηκε από το Φόρουμ για τις ΜΚΟ του 2011 για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ώστε θα πρέπει να λαμβάνεται επαρκώς αποτελεσματική δράση ε, επ' αυτών των θεμάτων όπως ζητούν οι ΜΚΟ ε, αφού γραζόμενοι αυτό το αίτημα και αυτές οι συστάσεις αυτό οδήγησε σε μια νέα εκστρατεία σε νέα διαβήματα τα οποία ε, ξεκίνησαν έναντι ε, χωρών που δεν έχουν ε, προσυπογράψει ή κυρώσει, επικυρώσει αυτές τις συμφωνίες και πρωτόκολλα. Και επιπρόσθετα, επειδή ο χρόνος πιέζει, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τις ΕΕ, για τις διαπραγματεύσεις, για μια συμφωνία για το εμπόριο, την εμπορία όπλων και οπλισμών και κατέστησαν σαφή την πεποίθησή του στα κράτη-μέλη ότι όταν υπάρχει σαφής κίνδυνο ε, να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους όπλα ή εξοπλισμοί για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την παραβίαση διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, τέτοιου είδους συναλλαγέ και πωλήσει όπλων θα πρέπει να απαγορεύονται υπό του όρου ε, τη. συνθήκη συνθήκης. Αυτή είναι κάποια από τους τρόπους, κάποια από τα μέσα που προσπαθεί να επηρεάσει τα πράγματα εφαρμόζοντας ε, τους, ε, τις κατευθυντήριες γραμμές για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ΕΕ. Ελπίζω να ικανοποίησα τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στην ειδική ε, κατάσταση στη Συρία. Ξέρετε αν αυτή η ομάδα εργασία του Συμβουλίου για το Διεθνέ Δίκαιο που θα έπρεπε να παρακολουθεί την κατάσταση που επικρατεί ε, έχουν συζητήσει την κατάσταση στη Συρία πρόσφατα. Και αν ναι, τι συνέχεια δόθηκε στη συζήτηση. για το αποτέλεσμα. The, ε, Απάντηση. Σύντομη απάντηση. Δεν γνωρίζω. Από ό,τι γνωρίζω από την εντολή που δόθηκε όμως στην ομάδα εργασίας, δεν είναι άμεση ευθύνη να συζητήσει γεωγραφικές καταστάσεις. αυτό το κάνουν οι αρμόδιες ομάδες εργασίας. Πρέπει να ελέγξω για να είμαι βέβαιος. Πρόεδρος, δεν είμαι ειδική, όμως οι εμπειρογνώμονές μου μου λένε ότι έχουν καθήκον να παρακολουθούν καταστάσεις όπου εκεί που μπορεί να ισχύει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προτείνουν λύσεις. Δίνω το λόγο στον David Νίκολς από τη Διεθνή Αμνηστία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την εφαρμογή, μάλλον μην εφαρμογή, ε, των κατευθυντήριων γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να συναγάγουμε μαθήματα για την όλη κατάσταση που επικρατεί στη Συρία. Όπω σωστά είπατε και όπω αναφέρθηκε και από τον εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η Διεθνής Αμνηστία μαζί με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις πώς οι κατευθύνες γραμμές για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν εφαρμόστηκαν όσο θα έπρεπε και είναι πολύ καλέ κατευθυντήρες γραμμές, σύντομες, εστιασμένες επί των δράσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Um, little, um, λοιπόν, Πρέπει να διαδοθούν οι γνώσεις ανάμεσα στους ε, φορείς για το πώς εφαρμόζονται. Και απ' έξω είχαμε λίγα στοιχεία ότι εφαρμόζονται. Και έτσι οδηγηθήκαμε να το θέσουμε σε βασικό θέμα προς στο φόρουμ του 2011 Ευρωπαϊκής Ενώσεως Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Θέλαμε να βρούμε λεπτομέρειες. Πώς εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και ποιος είναι υπεύθυνο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εφαρμογή του. Και να καταλήξουμε στις συστάσεις για να βελτιωθεί η εφαρμογή, η υλοποίησή τους. Στο φόρουμ των ΜΚΟ ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα. Είδαμε ότι δεν εφαρμόζονταν σωστά οι κατευθυντικές γραμμές. Κυρίως λόγω ελλείψης πολιτικής βούλησης των κρατών μελών. και επιμερισμός ευθυνών ήταν ασαφής για την υλοποίηση. Διάφοροι φορείς Ευρωπαϊκής Ενώσεως έπρεπε να ενεπλέκονται στον τομέα αυτό, αλλά όσο πιο πολλοί αναμειγνύονται, τόσο λιγότερα τα αποτελέσματα, λόγω ελήψεως σαφών ευθυνών. Τι άλλο ανακαλύψαμε. Ότι η διατύπωση, το κείμενο σε δηλώσει Ευρωπαϊκή Ενώσεως για το Διεθνέ Δίκαιο ε, ε, ήταν ασαφέστατη ανακριβής, ασαφής. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες ε, έπρεπε να συμμετέχουν περισσότερο στη διατύπωση. Και η γεωγραφική κατανομή ήταν ασαφής. Αναφερόταν διάφορες καταστάσεις σαφώς και άλλες καταστάσεις όχι, λόγω πολιτικής, έλλειψης πολιτικής βούλησης. Τέλος, ο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δεν ενσωματωνόταν στις δράσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως. όπως στρατηγικές κατά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν αναφερόταν, ούτε σε σχέδια δράσης, ούτε σε άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει. Λοιπόν, από το φόρουμ του 2011 καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Πέντε είναι τα βασικά. Πρώτον, το θεσμικό πρόβλημα, η περίπλοκη δομή και έλλειψη κατανομής ευθυνών έπρεπε να λυθεί αμέσως. Να υπάρχουν σαφείς ευθύνες, ποιος έχει ευθύνη γιατί και για να εφαρμόζονται καλύτερα οι κατευθυντικές γραμμές για το θησαυροπιστικό δίκαιο. Και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετείται όταν διαπιστώνονται παραβιάσει του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και να θέτει το θέμα αυτό σε πολιτικό διάλογο ή ουδήποτε επίπεδο. Και σε διάλογο σε διεθνή βήματα με τρίτε χώρε. Τρίτον, οι κατευθυντήριε γραμμέ έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Δεν αναφέρεται σαφώς οι κατευθυντές γραμμές η καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Λείπει αυτό από τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως για καταστάσεις σε διάφορες χώρες μετά από σειράξεις και συγκρούσεις. Θα έπρεπε όσον αφορά τι παραβιάσει να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις τρίτες χώρες. Έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια. Αυτό είναι το τέταρτο συμπέρασμα. Πέμπτον, θα έπρεπε να εφαρμόζεται η θέση της Ευρωπαϊκής όσον αφορά την εξαγωγή όπλων σε συνάρτηση με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και όσον αφορά να αναφέρεται αυτό και να λαμβάνεται υπόψη διαπραγματεύσει τη Ευρωπαϊκή Ενώση σε διεθνή βήματα για τι συνθήκε για του εξοπλισμού. Αυτά απέρευσαν όπω προανέφερα από το Φόρουμ του 2011. Έκτοτε, τι συνέβη. Όπω είπε σωστά εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία, στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στο σχέδιο δράσης αυτή η πτυχή αναφέρεται, αυτό που υθετήθηκε τον Ιούνιο, φανταστικό, υπέροχο. Λαμβάνεται υπόψη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ενώσης, λαμβάνεται υπόψη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωση για τα ανθρωπιστικά θέματα, το πλαίσιο αυτό για τις κατευθυντικές γραμμές Χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Οι βουλευτές πρέπει να δουν το κοντζού τι ακριβώς έχει αποφασίσει, ούτω ώστε τα αποφασιστέντα να εφαρμόζονται καλύτερα. Και οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να σωματωθούν σε θέματα όπως είναι οι στατικές για κάθε χώρα και τα σχέδια δράσης θα πρέπει να συναθριστούν όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι υπεύθυνοι ποικιλοτρόπως για το διεθνές δίκαιο. Εντός των διαφόρων φορέων που συζητούν και εντός των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Έγιναν βήματα πρόοδου. Όμως παραμένουν τρία αρκετά μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντηριών γραμμών. Θα αναφερθώ σε αυτά. Πρώτον, σχετίζεται και με το ερώτημά σας για τη Συρία. Δεν συζητούνται στο Συμβούλιο καθόλου οι καταστάσει διάφορε χώρε όσον αφορά το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν υπάρχει βήμα που να συζητείται η κατάσταση που επικρατεί σε διάφορε χώρε όσον αφορά το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα έπρεπε να συζητούνται στι γεωγραφικέ ομάδε εργασία του Συμβουλίου, όμω δεν γίνεται κάτι τέτοιο. δεν έχουν καν την, ε, την ε, γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη για να συζητήσουν περίπλοκες νομικές λεπτομέρειες. Όπως σωστά είπατε, αν δεν συζητούνται σε ομάδες εργασίας γεωγραφικές, στην Κοντζούρ θα έπρεπε να συζητούνται, ε, στην ομάδα εργασίας του Διεθνές Δίκαιο στον τομέα. Και από... Είπαν οι διάφοροι πρόεδροι της Κοντζούρ ότι δεν είναι στην εντολή που τους έχει δοθεί να συζητούνται ξεχωριστά χώρες. Άρα δεν συζητείται καθόλου το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στο Συμβούλιο και θα συμφωνούν όλοι ότι αυτό είναι ντροπή. Πρέπει να διορθωθεί. Και σαν Μίκιο θέλουμε κοινοβουλευτική υποστήριξη για αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, οι δηλώσει πορέων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνάδουν με αυτά που έτσι το διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε σχέση με διάφορες χώρες και με τη διατύπωση και τον τόνο. Καμιά φορά είναι καλή διατύπωση, καμιά φορά είναι πολύ αόριστη. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πούμε. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η διατύπωση και η έκφραση. Και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου επίσης. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου περνάνε από εξέταση νομικών στις πρωτεύουσες των χωρών. Οι δηλώσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν εξετάζονται νομικά δεν είναι κάποιος που καταλαβαίνει το διεθνές ε, ανθρωπιστικό δίκαιο που συντάσσει αυτές τις δηλώσεις. Τρίτον, πώς να βελτιωθεί η τεχνογνωσία εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης λέγουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε στρατηγικές για χώρες και διαδράσεις, σε διάλογο κλπ. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη. Ε, να, οι επιτόπου αντιπροσωπείς να ενημερώνουν το κέντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει αυτό άμα δεν υπάρχει εμπειρογνώμων που να ξέρει την κατάσταση και δεν κάνει τον έλεγχο εν πρώτης. Χρειάζονται περισσότεροι εμπειρογνώμονε να προσληφθούν να βασιζόμαστε στην εμπειρία των κρατών μελών και τεχνογνωσία, χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση. Αυτό θα μπορούσε να το θέσει σαν ε, ερώτηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει. Μπορώ να σταματήσω ή να αναφερθώ και στη Συρία, αν έχω χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Ναι, α, ωραία. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν. Κατάσταση στη Συρία. Και οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα. Είπαν ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία παραβιάσεως του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και μάλιστα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου που διαπιστώνονται στη Συρία. Το ανέφερε η Ερευνητική Επιτροπή και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως εμείς και η Human Rights Watch. περισσότερες γίνονται από την κυβέρνηση αλλά έκανα και εγκλήματα πολέμου και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης και παρόμοιες πράξεις. Ποια ήταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προσπάθησαν να οθήσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραπέμψει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την κατάσταση στη Συρία. Όπως είπατε όμως δεν υπάρχει πρώτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως πάνω σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή δεν ζητά να γίνει παραπομπή στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο γιατί ένα κράτο μέλο είναι αντίθετο. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την επόμενο, τον επόμενο μήνα να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαν ότι θα ήθελαν οι ευθύνε να αποδοθούν. Υπάρχει όμως μπλοκάρισμα, όπως είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλε δύο για να δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί στην κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει εμπάργο για τα όπλα στη Συρία. Έχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων παρέμεινε αυτό παρά το ότι ένα-δύο κράτη-μέλη είπαν ότι πρέπει να αρθεί το εμπάργο. Υπήρξε συμφωνία όμως να δοθεί μη ε, βοήθεια που δεν είναι ε, τεχνική βοήθεια στην αντιπολίτευση, όχι όπλα, όχι φωνικά όπλα, όχι φωνικά μέσα μάλλον θα πρέπει να γίνει εξολόγηση κινδύνου. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί για παραβίαση διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Όπως είπατε υπάρχει και κρίση ε, προσφύγων, πάνω από 620.000 πρόσφυγες έχουν φύγει από τη Συρία και πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας. Η Ιράκ, η Ορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία έχουν υποστεί το βάρος της κρίσης και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανταποκρίθηκαν μόνο μερικά στο πρόβλημα και απέρριψαν και επέστρεψαν πρόσφυγες. Δεν βοήθησαν τις γειτονικές χώρες να υποδεχθούν πρόσφυγες από τη Συρία, ούτε τις βοήθησαν τις χώρες να λύσουν τα εσωτερικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εισρωή προσφύγων. Αυτά είναι μερικά σχόλια που είχα, κυρία Πρόεδρε. Thank you, David. Now... ευχαριστούμε, David. Εσείς, κύριε Γκέρανς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ομολογήσω ότι αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα όταν συζητάμε τέτοια θέματα, διότι η τυπολογία των σειράξεων εξηγεί και την αδυναμία μας να κάνουμε κάτι. Και τη δεκαετία των 90 την ίδια συζήτηση κάναμε για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το Διεθνές Δίκαιο δεν επαρκούσε για να επιτρέψει μια εξωτερική επέμβαση. Και θυμάμαι τον Μπερνάχ Κουσνέχ που προσπαθούσε να υιοθετηθούν ε, τα ανθρωπιστικά δικαιώματα και πάντοτε αντιμετωπίζουμε και τώρα πάλι τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους φραγμούς. Κάποιες ε, προσωπικότητες ε, υπεράνω πάσης υποψίας, ο κ. Σουμαρούγκα παραδείγματο χάρη, ε, έκαναν προσπάθειες για να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο με τίτλο «Ευθύνη προστασίας». Έγινε η, ίδια ανάλυση και ακούγοντα τον κύριο Λάγκ, θυμήθηκα ότι ακριβώς την ίδια ανάλυση είχαμε κάνει στο πλαίσιο του εγγράφου «Ευθύνη προστασίας». Ακριβώς τις ίδιες αδυναμίες διαπιστώσαμε και για να, δείξουμε, να σας δείξω σε τι βαθμό ε, έχουμε πλήρη αδυναμία για τη Συρία, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και στο έγγραφο αυτό για την ευθύνη προστασίας. Αυτό που λέει είναι ότι ε, μπορούμε να παρέμβουμε αν ε, το πρόβλημα είναι σχετικό. Προφανώς μια επέμβαση έχει σχέση με το πρόβλημα. Δεύτερον, εάν τηρείται κάποια αναλογικότητα. Τρίτον, εάν ε, η παρέμβαση λύνει περισσότερα προβλήματα από όσα δημιουργεί. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι προτάσεις του εγγράφου ευθύνη προστασίας είχαν υιοθετηθεί, πάλι αδυναμία θα είχαμε για την κατάσταση στη Συρία. Διότι το να ε, εμπλακούμε στρατιωτικά σε μια τέτοια σύραξη δεν λύνει τα προβλήματα κάποια προβλήματα μπορεί να λύνει, αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα που παραμένουν θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα. Λοιπόν, καταδικάζουμε τα προβλήματα, αναζητούμε λύσεις και νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια προσπάθεια να βρούμε διάφορες λύσεις γύρω-γύρω από το πρόβλημα, ενώ παράλληλα ομολογούμε την αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε το ίδιο το πρόβλημα όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μεταξύ όλων των φορέων, όλων των θεσμικών φορέων, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την καλύτερη δουλειά. Η κυρία Γεωργίεβα κατάφερε να κάνει ό,τι μπορούσε, έφτασε πραγματικά στο όριο αυτών που μπορούσε να κάνει, λαμβανωμένων υπόψη των ε, δημοσιονομικών περιορισμών και των περιορισμών του διεθνούς δικαίου και το κατάφερε διότι ε, έχει την αναγνώριση των εμπλεκομένων στη σύραξη ως προς την αμεροληψία της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να δράσει στο πλαίσιο της σύραξη στη Συρία, όπως επίσης και στο Μάλι. Επομένως, ένα δίδαγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η αμεροληψία είναι το, ο απαράβατος όρος για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια τελευταία παρατήρηση εν είδη προτάσεως. Ο τύπος σύραξης που αντιμετωπίζουμε είναι μη διεθνής τύπος σύραξης. Η σύμβαση της Γενέβης εφαρμόζεται στις διεθνείς σειράξεις. Το διεθνές δίκαιο δηλαδή ε, είναι προετοιμασμένο για τέτοιου είδους συράξει διεθνείς. Για μη διεθνείς συμβάσεις δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα και αυτό πρέπει να το πούμε. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 λέγαμε ότι στη Ρουάντα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ένα μηχανισμό προειδοποίησης. Τι προειδοποίηση αφού όλοι τα ξέρανε. Όλοι ξέρανε τι συνέβαινε αλλά δεν είχαμε δυνατότητα παρέμβασης. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι η φρικτή κατάσταση την οποία διαπιστώνουμε ε, στις σφαγές που γίνονται στη Συρία και αλλού ε, απαιτεί ε, δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας. Θα πρέπει στην εκπαίδευση της αστυνομίας σε κάθε χώρα να εντάσσονται τέτοια ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και θα έπρεπε να απειλούνται με κατηγορίε εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας αν δεν τηρούν αυτό το διεθνέ δίκαιο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, δηλαδή να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε όλου του υπεύθυνου για την επιβολή τη τάξη μέσα σε μια χώρα. Θα πρέπει αυτοί να φροντίζουν να τηρούν και το διεθνέ δίκαιο και το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Και τελικά, αν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, αν ε, μια χώρα δεν ανταποκρίνεται στις ευθύνες που θα έπρεπε να αναλάβει, αν οι δομές της χώρας δεν ανταποκρίνονται, παραμένει η κοινωνία των πολιτών. Αναφέρατε την Ερυθρά ημισέλινο, που σε, που σε ορισμένες περιπτώσεις κάνει πολύ καλή δουλειά. Ίσως πρέπει να περιμένουμε, όπως είπατε, μέχρι το 2015 για την επόμενη διάσκεψη. Ε, ακούγεται κάπως γελίο, γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οργάνωση μια διάσκεψη μεταξύ τη Ερυθράς Σιμισελίνου και τη Διεθνού Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, ενισχύσουμε και την αμεροληψία και την δυνατότητα δράση. Στι περισσότερε από αυτέ τι χώρε υπάρχει και ερυθρά ημισέλινο, άρα υπάρχει σαφώ ένα πρόβλημα που πρέπει στο πλαίσιο ενό διαλόγου να επιληθεί. Και ξέρω ότι η Ελβετία και όσοι εκτελούν τις συμβάσεις της Γενέβης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Σύστημα κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτές είναι οι προτάσεις μου προς τον κύριο Λάγκ. Δεν ξέρω αν επιλύουν το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να παραμείνουμε με τα χέρια δεμένα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. κάθε φορά που αναφέρονται αυτά τα προβλήματα, το μόνο που διαπιστώνουμε είναι η αδυναμία μας. Αυτά λοιπόν είναι τα σχόλιά μου και σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους παρενέβησαν για τα όσα μας είπαν. Αληθεύει όπως είπε ο κ. Γκέρανς, ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα όλους μας. Μας αφορά όλους μας επειδή αφενός έχουμε τον πρέσβη της ε, Ελβετίας ε, και έκανε λόγο για το, το ανθρωπιστικό δίκαιο και από την άλλη πλευρά έχουμε πολύ λίγο προχωρήσει. Δεν έχουμε καθόλου προχωρήσει σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο. Όταν ακούγαμε τη Δευτέρα την κυρία Επίτροπο Γεωργίευα να κάνει λόγο για ε, την κατάσταση σε σχέση με τον προϋπολογισμό για το, τα, τις ανθρωπιστικές δράσεις που θα είναι μειωμένος κατά το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιτόπου παρατηρητές ε, που θα μπορούν να υποπτεύουν και να παρατηρούν την υλοποίηση των όρων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαιωμάτου και την συμμόρφωση και όλα αυτά με περιορισμένα κονδύλια. Εγώ είμαι υπέρμαχος φυσικά να συνεχίσουμε την προσπάθεια όπως αναφέρθηκε σε σχέση με αυτή την προσπάθεια. Έκανε λόγο και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διπλωματικής Δράσης και πρέπει να, στον πολιτικό μας λόγο να εισαγάγουμε την ε, συμμόρφωση με τις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Πρέπει να υπάρξουν όμως πηγές για την υλοποίηση, πηγές και ε, δυνατότητες για την υλοποίηση αυτή. Και εδώ θα ήθελα να προβληματιστώ κατά κάποιο τρόπο και ελπίζω να μην ε, ενοχλήσω καθόλου τον κύριο πρέσβη, τον κύριο πρέσβη της Ελβετίας. Πίσω από την μη σε πολλές περιπτώσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου βρίσκονται πολλά άλλα αίτια, πολλά βαθιά αίτια και που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως είναι το εμπόριο όπλων, το εμπόριο ανθρώπων, όπως είναι το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και πίσω από όλα αυτά πάλι υπάρχουν άλλα πολλά αίτια και αυτό πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη στη μάχη και στον αγώνα μας. Γι' αυτό δεν πετυχαίνουμε τα αποτελέσματα που μπορεί, πρέπει να είναι σε βάθος γιατί δεν καταλήγουμε στο βάθος των προβλημάτων και πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα και να δούμε αυτό σε βάθος. Μπορούμε να ζητούμε πολλά πράγματα αλλά δεν είμαστε πολλές φορές σε θέση ούτε να κάνουμε το σωστό πράγμα ούτε να ζητήσουμε τα αναγκαία. Στον πολιτικό διάλογο θα πρέπει να διατηρηθεί να αυξηθεί στο μέτρο που μπορείτε το, η συμμόρφωση και η ευθυγράμμιση με τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου και παρακαλώ όλοι μας, όλοι οι ευρωβουλευτές αυτού του σώματος Όλοι να είμαστε σε διάθεση και να μπορέσουμε όλοι να συνεργαστούμε και να συνεισφέρουμε. Όχι μόνο να υπάρξει κάποια διεθνή συνεργασία, όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια από πλευράς αυτού του Κοινοβουλίου να μην περικοπεί, να μην περικοπούν τα κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτές είναι οι αρχές που πρέπει να υπερασπιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, τουλάχιστον στην Επιτροπή Επιτροπή προς αυτό το στόχο και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουν αυτή την προσπάθεια προς αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας πιέσω να σας υποχρεώσω να μιλήσετε. Ποζωτά. Να πω κάτι. Δεν είχα δυστυχώς την τύχη να ακούσω τους ε, ομιλητές. Ε, δεν ε, θα ήθελα να πω κάτι λοιπόν. Ήμουν στη Συρία όμως και είδα αυτό το πρόβλημα, το παρακολούθησα από το 2004. Και πράγματι το χάσαμε το ραντεβού με τη Συρία. Δεν καταφέραμε να υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, δεν καταφέραμε για πολλούς λόγους και ποτέ δεν καταφέραμε να έχουμε έναν μοχλό θετικό επί των εξελίξεων στη Συρία και κάποια δεδομένη στιγμή θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχασε το τρένο και το ίδιο και η Συρία. Και αυτή η Συρία που χαρακτηριζόταν και εδώ έχω το ίδιο πρόβλημα όπως και με το, με το χάλι στο Ιράκ. Η Συρία αυτή είχε μια κοινωνία ε, μορφωμένη, συστήματα δημόσια που λειτουργούσαν με ένα καθεστώς ε, αστυνομικό απίστευτα περίπλοκο, κάτι που δεν παρουσιαζόταν ως δικτατορία, αλλά το αυταρχικό καθεστώς όσον αφορά την καταπίεση. Είχαμε αντιπολιτευόμενους όπως τον Γκυλό που μπορούσε να μιλήσει όσο μπορούσε και μετά ξαφνικά τον φυλακίζανε, τον βγάζανε από τη φυλακή κλπ. Ήταν ένα καθεστώς τρόμου. Παρόλα αυτά ε, υπήρχε, ήταν λαϊκό κράτος, ε, υπήρχε ανεξιθρησκεία φανταστική. Ε, υπήρχαν πολύ σημαντικά στοιχεία που τη διαφοροποιούσαν τη Συρία της άλλες χώρες. Ξαφνικά, μέσω μιας αραβικής άνοιξης που στην αρχή ε, υποστηριζόταν από του προσφυστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την νεολαία κλπ. που επαναστατούσαν κατά των αστυνομικών καθεστώτων. Πώ φτάσαμε σε αυτό τον πόλεμο, τον εμφύλιο, βλέπουμε να κατέβονται και άλλοι, Ιράν, Ρωσία κλπ. που δίσδυσαν όλοι αυτοί εκεί. Οι ε, λένε επιτίθεστε στο, στη Συρία, ε, αν επιτεθεί κανείς στη Συρία επιτίθεται κατά τη, του Ιράν, κατά της ε, Ρωσίας, γιατί είναι μέσα. Και έγινε κάτι που δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε, που δεν μοιάζει πλέον με τη Συρία εδώ, που είχαμε εδώ και μερικά χρόνια. Και λέμε ότι αν τα αγγίξουμε εκεί θα την αχτούν τα πάντα στον αέρα, ο Λίβανος είναι δίπλα κλπ. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν είναι επειδή είμαστε αδύναμοι, ε, θεμελιώς λέω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο κίνδυνος γενικής αναζωπήρωσης έκρηξης όταν έχουν ανακατευτεί όλη η Συρία θα είχαμε περισσότερη δυνατότητα δράσης. Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα που δεν υπάρχει παρά μόνο μια πολιτική λύση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει παρά μικρή δυνατότητα, άλλη δυνατότητα, λαμβάνοντα υπόψη τις δυνάμεις που είναι εντός της Συρίας και που παίζουν εκεί μέσα, η λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική η πολιτική χρειάζεται χρόνο κλπ. Και εν τω μεταξύ ο κόσμο προσπαθεί να ξεφύγει, ο κόσμο πεθαίνει, η επανάσταση δεν έχει το ίδιο πρόσωπο που είχε, ο πόλεμο μεταξύ θρησκειών πολλαπλασιάζεται, σιίτε κατά σουνητών κλπ. Ε, γίνεται κάτι που είναι σαν ατομική βόμβα. Η αδυναμία οφείλεται σε αυτό, δεν οφείλεται σε έλλειψη πρόβλεψης, δεν οφείλεται σε εμπόριο ναρκωτικών, οφείλεται για την ώρα στην διείσδυση όλων των δυνάμεων των περιοχών που έχουν διεισδύσει και στη Συρία. Προσπαθείτε να, να απαγορεύσετε υπερπτήσεις και κάνετε μια ελαφρά στρατιωτική παρέμβαση, μπαίνετε σε τεχνικούς Ρώσους, ε, επιτετραμένους Ρώσους κλπ. Είναι δραματικά αυτά τα πράγματα, αλλά ομολογώ ότι βλέπω πολιτική υστέρηση του είμαστε πολύ ήπιοι. Ε, δεν καταφέραμε να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία, με την Κίνα, να διαπραγματευτούμε ε, κάτι, ε, να ασκήσουμε τον Μπασάρ. Ο Μπασάρ δεν θα υποχωρήσει ποτέ. Θα βγει με τα πόδια μπροστά μόνο. Δεν είναι τρελός αιμοσταγής σαν τον Κατάφη, αλλά είναι ομός, βίος, ε, βιοπραγή, είναι πολύ βίος και δεν θα κουνηθεί. Όλος ο κόσμος το επιβεβαιώνει ότι τον ξέρανε. Αυτό είναι τρελός. Δεν είναι τόσο τρελός όπως ο Καντάφη, αλλά έχει τη δική του τρέλα, ιδιαίτερη τρέλα, και να προσπαθήσει κανείς να, το, να τον βάλει στην άκρη, να βάλει προσωρινή ε, κυβέρνηση και να τον παραμερίσει σιγά σιγά. Όλα αυτά συζητήθηκαν, συζητήθηκαν, αναφέρθηκαν, αλλά δεν υπάρχει παρά μόνο μία λύση. Μία λύση πολιτική. Και πολιτικός θα πρέπει να πλήξουμε και να ασκήσουμε πιέσεις. Αυτά ήθελα να πω. Λυπούμε, λυπούμε, λυπούμε που ήμουνα στον Κάρελ Μπίλτ δίπλα και δεν ήμουν παρούσα. Είναι γελίο που ζήτησα το λόγο, αλλά ήθελα να εκφράσω και εγώ την οργή μου ε, έναντι της αδυναμίας. Ε, λυπάμαι που δεν είχα δυνατότητα να σας ακούσω και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέρεν, ζητήσατε το λόγο. Μπορεί να είστε πολύ σύντομος, σας παρακαλώ ένα σχόλιο. Έχω και μια ερώτηση. Σχόλιο. Τακτικά μου συμβαίνει να ακούω το όνομά μου να σφαγιάζεται. Δεν είμαι. Γκέρινγκ, είμαι Γκέρινγκ. Γιατί σφάζεται το όνομά μου πολλέ φορέ στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο σε αυτέ τι περιστάσει που καταδικάζουμε όλα αυτά που ενσαρκώνει η προσωπικότητα του Γκέρινγκ. Ξέρω ότι εκείνοι που έχουν διαπράξει τη σφαγή του ονόματό μου το έκανα συνείδητα. Σα το λέω φιλικά. Δεν είναι ευχάριστο να επαναλαμβάνετε αυτή τη σφαγή του ονόματό μου. Λοιπόν, το ερώτημα. Σύμφωνο με αυτά που είπε η Βερονίκ Κάιζερ, αλλά έχω μια ερώτηση προ του υπερασπιστέ του διεθνού δικαίου, όπω είμαι και εγώ. Όπω βλέπετε εσεί και αντιλαμβάνεστε το δίκαιο, αν συνάδει το ότι δίνουμε όπλα στους ε, αντάρτες αυτού του συγκρούσεις. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι παραδίδονται παραδίδονται στα χέρια της κυβέρνησης αυτά. Θα δεχόσασταν να δώσουμε τελικά, ε, βλέποντας πόσο σοβία είναι η κυβέρνηση, να δίνουμε όπλα σε αυτούς που αντιτάσσονται στην κυβέρνηση. Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω το λόγο αν θέλετε να μιλήσετε. Ο κύριος ε, Νίκολς μπορεί να πάρει το λόγο πρώτος και μετά συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσω ε, από την τελευταία ερώτηση για το να εξοπλίσουμε την αντιπολίτευση. Δεν είμαι βέβαιος το τι χρειάζεται στη σύγκρουση. Χρειάζεται περισσότερα όπλα να μπουν στην όλη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει σαφείς κανόνες πότε μπορεί να απολύσει και πότε μπορεί να δώσει όπλα ε, και ε, διάφορα μέσα θανάτου, θανάτωσης δεν μπορεί να διευκολύνει όμως την παραβίαση διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή το διεθνές, ε, τα διεθνή θεμελιώδη δικαιώματα. Ούτε εμείς ούτε άλλοι, άλλες οργανώσεις έχουν δείγματα ότι παραβίαζαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και οι αντάρτες. Ή μάλλον έχουν παραβιάσει και αυτοί. Και εγκλήματα πολέμου και κατά Δεν είναι θέμα του να εξοπλίσει την αντιπολίτευση. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη αξιολόγηση κινδύνου από ό,τι έγινε. Περισσότερος διάλογος. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών που ανέφερα τη παραδιά. Ευχαριστώ, ο πρέσβη ο κύριο Λαό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας απαντήσω ή να σας συγχαρώ για την ανάλυση σας. Πολύ σωστή η κατάσταση που περιγράφατε κατά την άποψή μου είναι αυτή που επικρατεί. Είναι δυσκολότατο να κάνουμε κάτι και η χώρα μου πιστεύει ότι υπάρχει μόνο η πολιτική λύση, διότι είναι τέτοια απειρήτητα εκεί, ε, μπορεί ακόμα επιδεινωθεί. Ε, η λύση θα πρέπει να βρεθεί μέσω από μια πολιτική λύση, όσο και δύσκολη να είναι. Καταλαβαίνω, κύριε Γκέρενς, ότι εκνευρίζεστε, που δεν γίνεται τίποτα, τίποτα δεν συμβαίνει, καμία βελτίωση. Ο ρόλος μου εδώ, γι' αυτό ήρθα, είναι να υπερασπιστώ την εξής ιδέα. Υπάρχει ισχυρό διεθνές δίκαιο που δημιουργεί μια ισχυρή διεθνή νομολογία και έχει δυνατότητες. Και είναι καθήκον μας και καθήκον της Ελβετίας και το κάνουμε σε άμεση συνεργασία με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να κάνουμε ό,τι μπορούμε διπλωματικά, ούτω ώστε τελικά να αλλάξουμε τα δεδομένα. Τώρα, για να υπερασπιστώ ότι έγιναν λίγα μέχρι τώρα. Η δεκαετία του 90 μετά τον ψυχρό πόλεμο ήταν, αλλά ε, είχαμε προβλήματα εκείνη την περίοδο. Είχαμε και επιτυχίες. Σε στο Μπουρούντι, Ρουάντα, Σρεμπρενίτσα σε, φρικτές, σε φρικτά πλαίσια. Όσον αφορά την καταστολή και την αποφυγή τέτοιων, ε, είχαμε κάποια επιτυχία και την μακροπρόθεσμη εφαρμογή του νόμου μέσω της πρόληψης επανάληψης τέτοιων φαινομένων. Τώρα, θέλουμε να δράξουμε την ευκαιρία που υπάρχει να δούμε μήπως μέσω διαδικασίας διπλωματικής πολύ ευαίσθητης, διότι είναι πολύ ευαίσθητοι όλοι εκεί, να προωθήσουμε το θέμα. Ελπίζουμε ότι με νέα προσέγγιση Δηλαδή να μην έχουμε δεδομένες προτάσεις έτοιμες που δίνουμε, αλλά μαζί να ετοιμάζουμε διαδικασίες μέσω διαλόγου. Να βρούμε ενδεχόμενε λύσεις. Μέσω τέτοια διαδικασίας, με την πάροδο του χρόνου, το ξέρω, να σημειώσουμε πρόοδο. Τετραετία θέλουμε μεταξύ των δύο διεθνών διασκέψεων. Ε, του Ερυθρού Σταυρού και Τη ε, της Ερυθράς Ημισελίνου και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο και η πολιτική δεν είναι ικανοποιημένη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και όπως είπα, ποια είναι η ιδέα να δημιουργηθεί αυτή η διάσκεψη των χωρών που θα συνεδριάζουν κάθε χρόνο, ώστε να μην σταματάει πλέον η συζήτηση. Διότι αν κάθε χρόνο γίνεται μια διάσκεψη, η συζήτηση πριν και μετά ε, ε, διακόπτονται ε, συνεχίζεται, δεν, χάνονται από την οθόνη του ραντάρ. Δηλαδή παραμένει η συζήτηση στην οθόνη. Αν είναι το χρονικό διάστημα χάνεται. Ευχαριστώ πρέσβη κύριε Λάγκ. Έχουμε διερμηνία για πέντε λεπτά λέει η Πρόεδρος. Κύριε Ντεμπράουρ παρακαλώ είστε σύντομο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Τρει παρατηρήσει μόνο. Άκουσα προσεκτικά τα όσα ελέγχθησαν, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή μια ισχυρή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεκτική γλώσσα όσον αφορά την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Διαπιστώνω ότι για την περίπτωση που μας απασχολεί σήμερα, αν αναφερθούμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, η παράγραφος 8 δείχνει ότι έχουμε μία ισχυρή και συνεκτική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για την ατιμορρησία, μιλάμε για τις ευθένες, μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ακόμη και αν υπάρχουν ε, διστάμενες απόψεις. Αναφερόμεθα στην επιστολή της ε, κυβέρνησης της Ελβετίας, κύριε Πρέσβη. Τουλάχιστον υπάρχει μία στεναρή γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο οφείλουμε να χαιρετήσουμε. Όσον αφορά το θέμα των όπλων, δεν θα εκφέρω γνώμη, αλλά βλέποντας πώς διεξήχθη η συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο, και συμφωνώ απολύτω με τον συνάδελφο της, Διεθνούς όταν μίλησε για το θέμα της αξιολόγησης κινδύνων. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που πρέπει να σταθμίσουμε πριν εκφέρουμε γνώμη. Ε, όσον αφορά τον επίγοντα χαρακτήρα και την ανάγκη εξέβρεσης λύσης, βεβαίως η υπεύθυνη ανθρωπιστικής βοήθειας με όλους τους φορείς του επιτόπου ε, βρίσκονται σε απόγνωση όσον αφορά τις διαστάσεις της κρίσης σήμερα και όχι μόνο στη Συρία, κυρία Ντεκάιζερ, αλλά και στις γειτονικές χώρες, γιατί αυτή η κρίση επιβαρύνει σε τεράστιο βαθμό όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση και το Λίβανο και την Ιορδανία. Πέραν των πολιτικών δηλαδή πτυχών και αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο αποσταθεροποίησης για τις χώρες αυτές. Από την πλευρά της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει μία μόνη πολιτική λύση. Χρειάζεται μία ε, πολιτική λύση ε, που θα διαρκέσει, μία μακροπρόθεσμη πολιτική λύση και αυτό αυτή είναι η μόνη λύση που μπορεί να βρεθεί. Και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτής να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σουάν, δεν θέλετε και πάλι το λόγο. Ούτε εγώ θα λάβω το λόγο για να βγάλω συμπεράσματα. Ε, νομίζω ότι όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, ε, αλλά από τις ε, παρεμβάσεις που έγιναν καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία. Συζητούνται τα θέματα σε γεωγραφικά μεμονωμένο επίπεδο και νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε εμένα από τους ΔΕΚ και καλό θα ήταν να κάνουμε άλλη μια συνάντηση και να καλέσουμε και τον πρόεδρο της ομάδας του Συμβουλίου για το Διεθνές Δίκαιο για να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες λύσεις που θα είναι περισσότερο εφαρμόσιμες. Θα δώσω το λόγο στην Εύα τώρα, κυρία Ζολή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους, διότι είναι δραματική η κατάσταση που διαπιστώνουμε. Δεν τα καταφέραμε να παρεμβούμε στην Συρία και να ηρεμήσουμε την τρέλα που επικρατεί. Υπάρχουν 300.000 πρόσφυγοι, 60.000 νεκροί και παράλληλα τα κράτη-μέλη με τον εγωισμό τους μειώνουν τη συνεισφορά μας. Μειώνουν την αναπτυξιακή βοήθεια που θα ήταν η μοναδική βοήθεια που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε και να επηρεάσουμε κάτι. Και αυτό το βλέπουμε στο Μάλι. Και είναι πολύ ανησυχητικό το ότι μειώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες ε, και να μαχόμεθα όπου χρειάζεται για να πείσουμε τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να συμφωνήσουν για να στείλουν, παραδείγματο χάρη, τον Ασάντ στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μα και σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή σα σε αυτή τη σημερινή ακρόαση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ. Sorry, Swan, can you speak to me directly or you... Ε, κύριε Σβάν, έχετε κάποιο σχόλιο πριν κλείσουμε. Παρακαλώ. Δεν θεωρήσα ότι υπάρχει λόγος να λάβω το λόγο μέχρι ότου κάνατε τις ε, παρατηρήσεις σας. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αφήσω να πλανάτε η εντύπωση που δώσατε ότι υπάρχει αδιαφορία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, δεν υπάρχει αδιαφορία για το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι σε τέτοιου είδους συναντήσεις ε, γίνεται πάντοτε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις προσπαθειές της και συμφωνούμε με αυτές τις ε, παρενέσεις, αλλά θα ήθελα για τα πρακτικά να καταγραφεί ότι και βέβαια ε, είμαστε αφοσιωμένοι στο, ε, στο σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα ήθελα και προσωπικά να αναφέρω ότι όταν εγώ ήμουν υπεύθυνο χώρας πριν αναλάβω ευθύνες σε θεματικό επίπεδο είχαμε ετήσια εκπαίδευση για θέματα διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και είναι κάτι το οποίο διαπνέει το έργο μας και θα ήθελα να το καταστήσω σαφές για τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε και ξέρετε ότι θα μπει στα πρακτικά αυτό και θα παρακολουθήσουμε το θέμα.